Bien. Eh bien, nous allons... Euh, Συνάδελφοι, να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας. Θα δώσουμε το λόγο στους ε, διερμηνείς μας για μια ανακοίνωση που δεν θα σα ευνηδιάσει. Ο λόγος τους διερμηνείς Για 36η μέρα συνεχίζουμε την κινητοποίησή μας λόγω της ε, μονομερούς επιβολής συνθηκών εργασίας από τη διοίκηση. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε σήμερα να υπερβούμε το ωράριο που προβλέπεται για τη συνεδρίαση ως τις 6.30. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς μας που έχουν και αυτοί τα δικά τους, αλλά θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τη δουλειά μας απόψε το σήμερα το απόγευμα. Εδώ λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, την Κεζίνε Μάισνερ, για τι λιμενικέ καταστάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τα χαρά να αναφερθώ λοιπόν σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω πως ε, οι σημαντικότεροι συνάδελφοι, α το πούμε έτσι, και όλοι συζητητέ δηλαδή βρίσκονται όλοι εδώ. Ήδη έχουμε συζητήσει αυτό το ζήτημα και ε, χαίρομαι που θα ξανασυζητήσουμε αυτή την έκθεση, η οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και είπα ε, ήδη στην Επιτροπή ότι θα την. Ε, πρόκειται να τη συγχαρώ γιατί πραγματικά ε, αυτή η έκθεση ε, μας βρήκε σύμφωνος σε μεγάλο ε, μέρος ε, και έχουμε κάνει μόνο μικρές κάποιε λίγε προτάσει τροποποιήσεων και ε, τη ίδια θερμή υποδοχή έτυχε αυτή η πρόταση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Οπότε συνεργαζόμαστε μάλιστα και με την Επιτροπή Περιβάλλοντο, ε, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να αναμένει κανεί εύκολα, γιατί συχνά έχουμε κάποιε αντίθετε απόψει, αλλά πραγματικά αποτέλεσε έκπληξη, μου είπε και ο συνάδελφο από την Επιτροπή Περιβάλλοντο, ότι δεν μα ε, προκάλεσε πολλά παράπονα αυτή η έκθεση τη Επιτροπή. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά. Έρχομαι τώρα στα τη έκθεση. Νομίζω πω οι σκιώδει είχαν τη δυνατότητα αναγνώσω την έκθεση και την είχα συντάξει και στα αγγλικά ε, για να είναι αναγνώσιμη από όλου. Και υπάρχουν κάποιες τροποποίησεις τις οποίες προτείνω εγώ και νομίζω ε, πως και οι τροπολογίες ε, που θα υποβληθούν ακολουθούν την ίδια συλλογιστική. Καταρχήν το, το ζήτημα εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν λιμένες, ε, τα οποία ε, ενδεχομένω θα έπρεπε να εξαιρεθούν από, την, ε, από το πεδίο εφαρμογή. Για παράδειγμα έχουμε την Αυστρία η οποία έχει και την Προεδρία του Συμβουλίου αυτή την περίοδο που δεν διαθέτει τέτοιου είδου θαλάσσιου λιμένε. οπότε μήπω θα πρέπει να εξαιρεθεί. Το δεύτερο τώρα ζήτημα είναι το εξή. Σε ό,τι αφορά την ποντοπόρα ναυσιπλοεία, έχουμε τους κανόνες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, έτσι, του ΑΕΜΟ. Και οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι τώρα ότι θεωρούσα πως όσα έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης Μάρπολ ε, έχουν και την πτυχή της προστασίας του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό ε, δεν είναι ε, πάντοτε τελικά, δεν ισχύει πάντοτε διαπιστώνω σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα απόβλητα που απορρίπτονται στη θάλασσα ή την επεξεργασία των λιμάτων και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα όσα συμφωνούνται σε επίπεδο σύμβασης Μάρπολ, αλλά για παράδειγμα εμείς μπορούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη ισχύουν πολύ πολύ αυστηρότεροι κανόνε. Οπότε, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτά τα υψηλά επίπεδα ε, και σε διεθνέ επίπεδο. Άρα λοιπόν. Νομίζω πως αυτό το διαπιστώνουν και οι σκιώδες συζητητές. Στο κείμενό μου προσπαθώ να πιέσω την Επιτροπή ως προς το να είναι πιο φιλόδοξη σε ό,τι αφορά αυτή τη σύμβαση Μαρπόλ. Για παράδειγμα, σε μια συνεδρίαση που επίκειται της, ε, του ΑΕΜΟ, του Διεθνούς Αυτιλιακού Οργανισμού, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα αυτά τα αλλιευόμενα απορρίμματα, αυτό το fishing for litter. Ε, δεν είχε ληφθεί υπόψη μέχρι τώρα, αλλά πραγματικά είναι σημαντικό. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν ξεκινήσει, για παράδειγμα στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες, όπου ε, δηλαδή το, ε, σκεπτικό είναι το εξή. Όταν υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία ε, ε, πλέον για αλληλεία και τελικά παθητικά συλλέγουν και απορρίμματα, τότε θα πρέπει να λαμβάνουν μια αποζημίωση για την εκφόρτωση αυτών των απορριμμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αντιπαραγωγική η όλη ε, προσπάθεια. Από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα της, ε, του περιορισμού των ποσοτήτων, γιατί υπάρχει βέβαια ε, και το ζήτημα των λιμένων στους οποίους καταπλέουν τα πλοία. Δηλαδή υπάρχει αυτό το 100% του έμεσου τέλους, δηλαδή το ότι μπορεί ένα πλοίο να καταπλέει, να πληρώνει αυτό το τέλος και να εκπορτώνει όλα τα, τα, τα απορρίμματα που έχει. Αυτό βέβαια είναι, σημαντικό, είναι, είναι απλό ο σύστημα και αποτελεί ένα κίνητρο ε, για να ε, εκφορτώνει κανεί όλα τα απορρίμματα του και τα λίμματα του στο λιμένα και όχι ακριβώ στην ανοιχτή θάλασσα. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, υπάρχουν κάποια λίγα, για παράδειγμα, υπολείμματα φορτίου ω απορρίμματα, ενώ υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία φέρουν πολύ υψηλή ποσότητα απορρίμματων δεν μπορούμε να λέμε με 100% καταβολή αυτού του έμεσου τέλους φάπαξ ε, ε, καλύπτονται τα πάντα σε ό,τι αφορά την ποσότητα των ε, απορριμμάτων. Τώρα ένα ακόμα ζήτημα το οποίο συζητείται αυτή την περίοδο και γνωρίζω προς τα που κινείται και το Συμβούλιο και το τι έχει προτείνει η Επίτροπη είναι ε, το κατά πόσο θα πρέπει κανεί να εκφορτώσει όλα αυτά τα απορρίμματα προτού εγκαταλείψει το τελευταίο λιμένα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για παράδειγμα, θα μπορούσε κανεί ε, να αναφέρει ένα παράδειγμα όπου ο τελευταίο λιμένα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ένα πολύ μικρό ε, λιμένας, ο οποίο για παράδειγμα θα είχε πολύ μεγάλα προβλήματα διαχείριση ενώ ο επόμενο λιμένας θα ήταν ένας μεγάλος. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τώρα και θα είχε τη δυνατότητα να λάβει περισσότερα απορρίμματα. Άρα λοιπόν ε, καλό είναι λοιπόν να προβλέψουμε τέτοιε δυσκολίε έτσι ώστε να γίνεται η ε, εκφόρτωση των απορριμμάτων ε, με το σωστό τρόπο στου λιμένε. Οπότε δεν πρέπει να είναι απόλυτο απόλυτος ο κανόνας σε ό,τι αφορά την εκφόρτωση όλων των απορριμμάτων εντός ε, λιμένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση Θα μπορούσε δηλαδή να προβλεφθεί και κάποια εξαίρεση. Από εκεί και μετά... Εγώ θα βρεθώ σε κανένα δυο λιμένες κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού διαλύματο, οπότε ε, ίσως θα έχω τη δυνατότητα να δω τι συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο διαθέτουν τι απαραίτητε εγκαταστάσει εκεί. Ε, τα, τα, τα λιμάνια. Για παράδειγμα, στο το Αμβούργο βρίσκεται ε, κοντά μου και έχει τα πάντα που εγκαταστάσει. Ενώ υπάρχουν άλλα μικρότερα λιμάνια τα οποία δεν έχουν τα πάντα, δεν έχουν καν αυτοματοποιημένα συστήματα. τα οποία για παράδειγμα δεν έχουν το, τα, κατάλληλα συστήματα σε ό,τι αφορά την έκδοση των σχετικών εγγράφων, άλλα δεν έχουν τις, αυτό ισχύει στον Βασίλειο, αλλά δεν έχουν τι κατάλληλε εγκαταστάσει για την παραλαβή των ε, απορριμμάτων. Και από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα της, ε, του διαχωρισμού των ε, αποβλήτων. Δηλαδή, ε, πλοία στα οποία ο διαχωρισμός γίνεται ήδη στο ίδιο το πλοίο, ενώ άλλες περιπτώσεις όπου πραγματικά όλα εκφορτώνονται από κοινού, το οποίο δημιουργεί με τη σειρά το περισσότερο πρόβλημα. Και κάτι ακόμα το οποίο μας απασχολεί όλους από κοινού είναι αυτές οι πλυντρίδες ανοιχτού βρόχου, αυτά τα, τα, τα scrubbers όπως λέγονται, ε, στην ε, Βαλτική, όπου ε, πάντοτε αναφερόταν ότι γίνεται αυτή η επεξεργασία του σκράμπινγκ και στη συνέχεια αυτά τα λίματα που προκύπτουν είναι καθαρά. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. δηλαδή, θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιούμε τους, τους, τα scrubbers, πράγματι, αυτές τις πλυντρίδες, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει Ε, να δούμε κατά πόσο θα συνεχίζεται να, επιτρέπει, να επιτρέπεται ή όχι η απελευθέρωση αυτών των λιματών ε, στη θάλασσα. Για τα παράδειγμα, στο Βέλιο ή στην ε, Γερμανία δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Σε άλλα κράτη-μέλη επιτρέπεται. Οπότε αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα κάνουμε ε, είμαι βέβαια ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία στο πλαίσιο αυτή τη ε, βουλευτική ακόμα περίοδου για να επιτύχουμε πιο καθαρέ ε, θάλασσε και με λιμάνια τα οποία θα λειτουργούν έβρισμα σε σχέση με αυτά τα απόβλητα. Αναμένω με ενδιαφέρον την συνεργασία που θα έχουμε με τους εσκιώδες συζητητέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε και τους σκιώδεις για το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας παρουσιάσατε, μας προτείνετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ γιατί από τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε εδώ στην Επιτροπή νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία για την πρόταση που μας υπέβαλε σήμερα. Νομίζω ότι αυτά που είπατε καλύπτουν και κάποιες από τις τροπολογίες στην 20, παραδείγματο χάρη. Νομίζω ότι η θετική σας πρόταση εδώ αναγνωρίζει ότι όλα τα πλοία δεν θα πρέπει να ξεφορτώσουν όλα τους τα απόβλητα πριν αποπλέψουν από το τελευταίο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό και πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει να κάνουμε. Είναι κάτι ιδιαίτερα για χώρες που βρίσκονται, αν θέλετε, έξω ή στα άκρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα εξωτερικά σύνορα και είναι λογικό. Είτε για μικρότερα λιμάνια, λιμάνια με λιγότερη κυκλοφορία πλοίων, θα πρέπει κάποιες από αυτές τις προτάσεις να μην ισχύουν υποχρεωτικά. Αυτό προτείνουμε στην τροπολογία 16. Νομίζω ότι αυτό που είπατε είναι πολύ λογικό. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διευθετήσουμε αυτές τις προτάσεις για να μπορούν να ανταποκριθούν και στις δυνατότητες των μικρών λιμανιών. Πολλές χώρες δεν διαθέτουν μεγάλα λιμάνια που να έχουν τις εγκαταστάσεις αυτές. Η κυρία Μάσνερ, αναφερθήκατε επίσης και σε θέματα... και των εξοπλισμών των μηχανημάτων αυτών που συλλέγουν τα απόβλητα, τα λευτικά αυτά μηχανήματα και εργαλεία. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε εδώ να ζητήσουμε να επομισθούν το βάρος αυτό οι αλίες. Θα πρέπει μέσω των ε, μηχανισμών χρηματοδότησης που διαθέτουμε να καλυφθεί το ε, έξοδο αυτό και βεβαίως να κάνουμε ό,τι γίνεται έτσι ώστε να μην συνεχιστεί η απόρριψη αυτών των αποβλήτων στη θάλασσα. Τώρα, αναφερθήκατε επίσης και στο θέμα της ε, θα πρέπει να προβλεφθεί και το θέμα των ε, μικρών διαδρομών κοντά στις ακτές, ε, της προτάσεις που κάνετε εδώ για τα τέλη νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να τις ξαναδούμε λίγο, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική ταξινόμηση των τελών. Βεβαίως, όλη η προσπάθεια είναι να σταματήσει η απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα με κάθε τρόπο, με επιβολή προστήμων, αλλά και με την ε, ύπαρξη κινήτρων ίσως εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο και τις διαδρομές ε, μεταξύ των λιμανιών και την κατανομή, αν θέλετε, της, ε, των ποσοτήτων στα μεγάλα και στα μικρότερα λιμάνια. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Επιτροπή προτείνει εδώ 100% έμεσο τέλος αυτό είναι μια τροποποίηση στον κανονισμό του IMO και ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε τι ακριβώς προτείνει εδώ η Επιτροπή. Γιατί η θέση του Κοινοβουλίου για αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί. Στην τροπολογία 10 θα πρέπει εδώ να ξαναδούμε λίγο την πρόταση αυτή γιατί πιστεύω ότι ο κανονισμός προβλέπει πολύ αυστηρούς κανόνες, άκαμπτους κανόνες όσον αφορά την καύση αποβλήτων. Θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι εδώ δεν παραβιάζονται κάποιοι άλλοι κανόνες ε, ναυτικού δικαίου. Είναι λίγο συγκεχημένες εδώ οι ορολογίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε ακριβώς τι ε, προβλέπεται για την καύση να δούμε τα διάφορα κανονιστικά κείμενα έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση. Συμφωνούμε επίσης και με την τροπολογία για την πράσινη ναυτιλία, green shipping. Παραθέτεται εδώ στο κείμενο μάλιστα και τα παραρτήματα της σύμβασης Marpol. με σκοπό να περιοριστούν και οι ποσότητες των σκουπιδιών των αποβλήτων που ξεφορτώνονται στα λιμάνια. Χαίρομαι ε, με αυτό που είπατε ότι θα συνεχίσετε να επεξεργάσετε το κείμενο του το καλοκαίρι, θα επισκεφτείτε και κάποια λιμάνια. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλοι εμείς που έχουμε εμπειρία να κάνουμε το ίδιο και με μεγάλη χαρά στην πρώτη μας συνάντηση το Σεπτέμβριο οι σκιώδες εισηγητές θα ξαναδούμε τις προτάσεις της Επιτροπής όταν θα έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι προτείνει η Επιτροπή. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Η κυρία Σαπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, την Κεζίνε, Αυτά που είπε είναι κέρια σημασία. Ξεκινήσαμε από ένα σχέδιο πρόταση τη Επιτροπή που ε, ήταν ε, Καλό, θα έχουμε βέβαια συζητήσει έπειτα και με του ε, σκιώδει εισηγητέ, θα έχουμε και περαιτέρω διαπραγματεύσει και σημείο σα είπε, είναι. Ε, δίκιο έχει τα περισσότερα, αλλά μπορούμε να έχουμε περαιτέρω συζήτηση και να δούμε συμβαστική λύση για τα εξή σημεία. Βεβαίω και εγώ θα υποβάλω τροπολογίε, αλλά νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να τα αποσαφηνίσουμε. Α μα τα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι, αλλά για παράδειγμα δεν έχουμε ακόμη ορισμό του green shipping, της οικολογικής ναυτιλίας, της πράσινης ε, ναυτιλίας. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι τα είδη σκαφών, οι κατηγορίες σκαφών που μπορούν να επωφεληθούν από όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε μαζί με την εισηγήτρια για να συνδυαστούν και οι τροπολογίες μας σχετικά. Έπειτα, δεν το είδα στι συμβαστικέ. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να βρούμε λύση. Δεδομένου ότι η ρήπανση εξαιτία των αποβλήτων που αδειάζονται, ε, αποτίθενται στον ε, Ρήνο, στο Δούναβη τελικά, ας πούμε από το Δούναβι, καταλήγουν ε, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό βλάπτει τα οικοσυστήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν πρέπει να ε, επεκταθεί ο κανονισμός και για τα λιμάνια της εσωτερικής ναυσιπλοείας των ποταμών που καταλήγουν σε κάποια θάλασσα. Θα πρέπει με κάθε τίμημα να αποφύγουμε τη ρήπανση, ακόμη και για τα ποτάμια. Έπειτα, μια άλλη ερώτηση που τέθηκε είναι γιατί να μην πληρώνει κανείς ανάλογα με τον όγκο το μέγεθος των αποβλήτων. Καταλαβαίνω αυτό που λέει η Συγγετρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν ε, θα είναι καλό να εκφορτώνουν τα απορρίμματά τους και τα απόβλητα στη θάλασσα για να γλιτώσουν ε, με μικρότερο όγκο τα πρόστιμα. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων των αποβλήτων. Όταν ε, μια κατηγορία ε, καταλήγει στην παραγωγή περισσότερων απορριμμάτων, θα πρέπει να την ε, αντιδιαστέλουμε από μια άλλη που παράγει λιγότερα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια σαφή διασύνδεση μεταξύ του όγκου των αποβλήτων από τη μία και τη πληρωμή ε, προστίμου που επιβάλλεται από την άλλη. Και μια άλλη πρόταση που μου φαίνεται ε, απαραίτητη για τα έντυπα εγγραφής θα πρέπει στην ανάλογη στήλη να αναφέρεται και ένας κωδικός ευρωπαϊκός, ο κωδικός για τα απόβλητα. Το συζήτησαμε με τις λιμενικές αρχές και δεν είναι εναντίον αυτής της ιδέας. Ε, θα πρέπει λοιπόν δίπλα στο κομμάτι που λέει ε, απόβλητα, καλό θα ήταν να υπάρχει και ένα κωδικός ευρωπαϊκός για το είδος του αποβλήτου, ε, να προβλεφθεί στα τυποποιημένα έντυπα βάσει του παραρτήματο 2. Και βεβαίω ε, κάποιες τροπολογίες που είναι ιδιαίτερα, ε, με βρίσκουν ιδιαίτερα σύμφωνοι, όπως με την τροπολογία 10. Εκεί προσπάθησες, Γκεζίνα, Γκεζίνε, να εξηγήσει τι είναι τα συγκεκριμένα απόβλητα ή στο, ε, στην τροπολογία 21. Και αυτή μου αρέσει πολύ. Είναι μια τροπολογία που δεν θα τη διαβάσω τώρα, αλλά θέλω να την αναφέρω. Και η 23, επίσης πολύ καλή τροπολογία, εάν ένα σκάφος χρησιμοποιείται για σύντομη απόσταση ναυσιπλοεία, μειώνεται η συμβολή του. Θα πρέπει να δούμε επίσης και το κατά πόσον ε, είναι επικίνδυνου χαρακτήρα τα απόβλητα, ε, μάλλον ποια είναι η επικινδυνότητά τους. Επίσης η τροπολογία 28 και 24. Υπάρχει μια προσθήκη εδώ. Προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, επιβάλλει κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει να ισχύσει το παράρτημα 5 της Σύμβασης Μάρπολ. Ε, και ε, εν τέλει να διευκρινίσω ότι θεωρώ όταν την επόμενη φορά θα συναντηθούν οι σκιώδεις εισηγητές η προθεσμία που έχει η υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2020 δεν είναι αρκετό χρονικό διάστημα εδώ είμαστε ήδη στα μέσα του 2018. Εγώ αυτό που προτείνω και ελπίζω να εισακουστεί είναι να δώσουμε ένα χρόνο παράταση, 2021 να πούμε. Δεν μπορούμε να προβλέπουμε προθεσμίες που είναι τελείως ε, μη ρεαλιστικές. Θα πιέσουμε κάποια κράτη-μέλη να δράσουν, να αναλάβουν δράση, θα βιαστούν και θα τα κάνουν θάλασσα. Μόνο και μόνο γιατί φοβούνται την προθεσμία. Μήπω και δεν τηρήσουν την προθεσμία. Αυτά είχα να πω. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλου του άλλου συναδέλφου, του του εισηγητέ και ελπίζω ότι ξεκινώντα από μια καλή λύση βάσει τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε κάτι ακόμα καλύτερο να προτείνουμε από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κυρία Γκραπίνη. Ο κύριο Βαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή την πρόταση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή και για το περιβάλλον, για τη βιωσιμότητα και νομίζω ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας παρακαλώ πολύ. Ας είμαστε λοιπόν προληπτική στη δράση μας. Δηλαδή, λιγότερες συσκευασίες. Μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να μειώσουμε τις συσκευασίες. Έχω την εντύπωση παρόλα αυτά ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία στην Επιτροπή μας και όσον αφορά το μάζεμα, την περισυλλογή των αποβλήτων, fishing for litter, όπως το λέμε, είναι μια πρακτική που βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να υπάρχουν αλλιευτικοί στόλοι οι οποίοι να έχουν μία δράση πολύ συγκεκριμένα για την συλλογή των ε, αποβλήτων υπάρχουν απόβλητα και στα βάθη των θαλασσών αλλά και που επιπλέον και θα πρέπει αυτό να είναι η κυρία δραστηριότητα για κάποιες συγκεκριμένες ημέρες του αλληλευτικού στόλου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να προσθέσω τα εξής. Ο δεσμευτικός χαρακτήρας αυτών των νομοθετικών προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να δημιουργούμε νομοθεσία. Είμαστε πολύ λιγότερο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα αυτών όλων των κειμένων και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν την τήρησή τους. Και βεβαίως ο ΑΙΜΟ, ο Διεθνής Οργανισμός ε, για την αυτιλία θα πρέπει εδώ να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο και την επιτήρηση. Στη χώρα μου, στην Ολλανδία, υπάρχει ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό δίκτυο συλλογής των αποβλήτων στη θάλασσα. Και θα πρέπει αυτό το μοντέλο, αυτό το δίκτυο να επικρατήσει και σε άλλες χώρες. Τα περισσότερα κράτη-μέλη σήμερα δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ε, έμεσα κάνουν ό,τι μπορούν αλλά αφού όλοι υπογράψαμε στην Συμφωνία των Παρισιών, αφού όλοι συμφωνούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για το κλίμα, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα των αποβλήτων στη θάλασσα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τα απομακρυσμένα λιμάνια, τα περιφερειακά λεγόμενα λιμάνια. Αναφέρονται αυτά στην έκθεση 18 και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την στήριξη. Όσον αφορά τώρα τα τέλη και τις έμεσες επιστροφές, σίγουρα, σίγουρα θα υπάρξουν πλοία τα οποία θα μεταφέρουν πολύ περισσότερα απόβλητα. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά ε, τις αποζημιώσεις για απόβλητα τα οποία θα ονόμαζα απόβλητα τα οποία ουσιαστικά ρίχνονται στη θάλασσα για να ουσιαστικά αποζημιωθεί η συλλογή τους εκ των υστέρων. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε καταρχήν είναι να επιβληθούν αυστηρότατες κυρώσεις σε αυτούς που μολύνουν Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέιλορ έχει το λόγο. I thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κεσίνα για τη δουλειά που έχει κάνει σε σχέση με αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, που πραγματικά θεωρώ πως αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη αρχή. Ε, χαιρόμαστε που βλέπουμε ε, πως ε, βλέπουμε να περιλαμβάνονται εδώ ε, μια σειρά από διαφορετικές επιγές αποβλήτων και επίσης και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυτά τα τέλη. Αυτή η αναφορά τώρα που γίνεται στην ασπλοεία μικρών αποστάσεων είναι ευπρόσδεκτη παρότι δεν είναι εύκολο να προφερθεί αλλά σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να περιληφθεί στην τελική έκθεση. Επίσης, αυτή η απαγόρευση της ε, απελευθέρωση στη θάλασσα όλων των ειδών απόβλητα, όλα τα, ε, δηλαδή από ρήματα ή υγρά, ε, η απο φορτια η η λυση για παράδειγμα από σκράμπερς όλα αυτά είναι ε, ε, θετικά ειδικότερα στο πλαίσιο ενός συστήματος το οποίο παρέχει κίνητρα για την εκφόρτωση αποβλήτων στα λιμάνια όπου αυτό είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη και αυστηρότερη εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών και εμείς θα προσπαθήσουμε να υπάρχει επιβολή κυρώσεων και προκειμένου η συμμόρφωση να λαμβάνει χώρα με βάση τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ε, διεθνώς σε ό,τι αφορά και την ε, διατήρηση της ε, βιοποικιλότητας και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Σύμβασης των Παρισιών. Και κάτι ακόμα που θα ήθελα να ακούσω, η ΕΜΣΑ δηλαδή ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, δεν θα μπορούσε να αναλάβει εδώ μία αρμοδιότητα συμπληρωματική σε σχέση με αυτό τον τομέα. Ευχαριστούμε πάντως την Επιτροπή για αυτή την πρόταση και την ευχαριστούμε για, ε, όπως ε, είπαμε, μια πολλά υποσχόμενη πρόταση από την πλευρά της ε, συναδέλφου ε, Gonzalez. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοντζάλες, θα ήθελα να καλωσορίσω την ομάδα του κυρίου Κράμερ. 30 άτομα που βρίσκονται εδώ στην αίθουσα και παρακολουθούν, η οποία είναι από το European Turning Center for Railways. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Σήμερα το απόγευμα δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για τους σιδηροδρόμους, μάλλον θα μιλήσουμε για τις θαλάσσιες μεταφορές. Voilà. Madame González, maintenant c'est à vous. Querida González. Muchas gracias, Presidenta. Pues aprovecho para saludar también al grupo y... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω και εγώ την ομάδα επισκεπτών του κυρίου Κράμερ. Το γνωρίζετε, είμαστε υπέρμαχοι των κρατικών σιδηροδρόμων ελπίζω να τις προωθήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο μέλλον. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ για την εξαιρετική της δουλειά σε αυτό το θέμα. Ε, είναι στο σωστό δρόμο και νομίζω ότι πολύ σωστά μας έχει ρυθμίσει την πορεία προς τον σωστό στόχο. Για αυτό το σειρμό μέτρων ε, υπάρχει μια σειρά από πράγματα που θα πρέπει να ε, τα δούμε πιο πρακτικά. Όταν λέμε τα μικρά λιμάνια ή τα περιφερειακά λιμάνια μπορούν να εξαιρεθούν. Τι θα πει αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάζουμε, να είμαστε προθύστεροι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας πει τι σκέφτεται, τι άποψη έχει για τα μακρινά λιμάνια πριν αρχίσουμε να μιλάμε για ε, εξαιρέσεις. Ε, μετά για την ε, ακτοπλοεία μικρών αποστάσεων. Ε, εκεί που θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερο κόστος. Οι τιμέ να είναι λίγο περιορισμένες. Επιμένω, τι θα πει αυτό, τι θα πει σύντομη απόσταση, πόσα χιλιόμετρα. Ε, μιλάμε για το καμποτάζ στη θάλασσα. Μιλάμε για συγκεκριμένες ε, επιχειρήσεις μεταφορών. Νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία χρήζουν περισσότερη διευκρίνηση. Επίσης, θέλω να επισημάνω και είχα την ευκαιρία να το πω και προηγουμένως, Πρέπει να έχουμε κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση τέλο πάντων για όλο το προσωπικό, όχι μόνο για όσους διαχειρίζονται τα απόβλητα, για το σύνολο όσων εργάζονται στις λιμενικέ εγκαταστάσεις, για όλους τους λιμανεργάτες. Είναι πολλέ οι λιμενικέ υπηρεσίε που μπορεί να επηρεαστούν από την αποκομιδή των απορρίτων. Ε, μετά, όταν μιλάμε για επιθεώρηση, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιε επιθεωρήσει απρόβλεπτες, τυχαίες, για να υπάρξει αποτελεσματικότητα ε, των ελέγχων. Και όταν μιλάμε για κυρώσεις, για πρόστιμα, θα πρέπει να είμαστε κάπως ε, ακριβείς στο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή να είναι σαφές ότι πρόκειται για δίκαιο κατά της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτές είναι μερικές από τις προτάσεις μου και πάλι ευχαριστώ την Κεζίνη, ευχαριστώ κυρία Μάισνερ και ε, εποφελούμε για να σας ευχηθώ και καλές διακοπές το ίδιο και στους Γερμανείς μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε κυρία Γκοντζάλες. Κυρία Μπελμπάο Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Γκεζίνε. Ευχαριστώ για την εξαιρετική σου δουλειά. Ε, ξέρετε ότι στην Επιτροπή Ελίας Είχαμε κοιτάξει τα αλλιευτικά σκάφη και τα ψυχογωγικά να μην ε, ε, συμπεριλαμβάνονται. Αλλά ξέρετε ότι κάποιες φορές κάποια δίχτυα ε, δεν είναι, ε, ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι αυτά η βασική πηγή ρήπανσης, είναι τα πλαστικά και δεν προκύπτουν από τα αλλιευτικά, δεν τα πετάνε τα, οι βάρκε που ψαρεύουν. Είναι μάλιστα πολλοί αυτοί που κάνουν προσπάθεια δια, διαλογή των πλαστικών ε, στο καράβι του, στο, στο σκάφο του. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε διάκριση μεταξύ των σκαφών που πάνε για αλεία ε, οργανωμένα και κάποιου που έχουν πάει για σκοπού ψυχαγωγικού, μια στι τόσε. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε όλου όμω για την αποκομιδή των απορρίτων. Απορρίτων που μπορεί να τυχαία να πιαστούν στα δίχτυα. Είναι πολλές οι αλλιευτικές ε, περίοδοι και τα ταξίδια για αλλία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε μεταξύ των αλλιών που ανήκουν στη μία στην άλλη κατηγορία και στα διάφορα λιμάνια υπάρχουν ε, σχετικές διαφορές δεδομένων των διαφορών στις ε, διαστάσεις κάποιων λιμένων. Κάποιοι δεν έχουν ε, συγκεκριμένα ε, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αλλά συνεργαζόμενοι με άλλα κοντινά λιμάνια μπορούν να κάνουν σωστή ε, συλλογή των απορρίτων και μετά το σωστό, τη σωστή διαλογή. Για τα απομακρυσμένα λιμάνια έχουμε υποβάλει κάποια σχετική τροπολογία. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και εξόχως απόκεντρες περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι χρηματοδότηση χρειάζεται για, την, ε, τον εξοπλισμό των λιμανιών αυτών. Είναι εξόχως απόκεντρα. Είναι σε ιδιαίτερα δυσχερή γεωγραφική θέση. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε πλατφόρμε σε συγκεκριμένα σημεία. Και πολλά από αυτά τα λιμάνια προσελκύουν και πολλού τουρίστε. Από μια άλλη άποψη λοιπόν, η ανάπτυξή τους βασίζεται στην ανακύκλωση με την κυκλική οικονομία ως προτεραιότητα. Το, αυτό ας πούμε ισχύει για τις Κανάριες νήσους και ε, για τέτοια νησιά θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κανόνες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε δραστηριότητες, σε οργάνωση της ανακύκλωσης βάσει της κυκλικής οικονομίας και για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Νομίζω ότι και εκεί τα λιμάνια αυτά θα πρέπει να ασχολούνται και με τις πηγές της μόλυνσης. Όσο για την προθεσμία της υλοποίηση, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν θα γκρίνουμε το κείμενό μας, να ξέρουμε ότι μπορεί και να ε, προλάβουμε. Και για τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες έχουν τις αρμοδιότητες αυτές ε, θα καθορίσουν τα προγράμματα διαχείρισης και αποκομιδής. Δεν μπορούμε λοιπόν να διοργανώσουμε ένα τέτοιο σύστημα για τα απορρίμματα κατά απόφλητα, αν δεν λάβουμε υπόψη μας στις αρχές τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Μεταφορών από την Επιτροπή Αλίας για να ε, επιτύχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Για ένα λεπτό ο κύριος Βαντενκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μία παρατήρηση έχω και μία ερώτηση. Πρέπει να σας πω ότι κάπως ανησυχώ όταν μιλάμε για μικρά λιμάνια και για μικρά σκάφη. Υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό με ανησυχεί, για τα μικρά σκάφη, τα οποία νομίζουν ότι είναι αδύνατο να ενσωματωθούν σε αυτούς τους κανονισμούς. Συνήθως όμως ξεχνάμε ότι μπορεί κάποιος να είναι μικρός αλλά να είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός, όπως παραδείγματος χάρη το Ντουμπρόβνικ. Η οδηγία, ναι, περί οδηγίας πρόκειται, αν λάβει υπόψη της και όλα τα στοιχεία που αφορούν το τουρισμό, θα μπορούσε να ενσωματώσει πολύ περισσότερα σκάφη που θα αφορούν και τα λιμάνια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ενσωματώνονται αυτά, ναι ή όχι στην πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βαντεκάμ και τώρα θα στραφώ προς την Επιτροπή. Βλέπετε ότι η έκθεση αυτή, η έκθεση της κυρίας Μάισνερ, προκαλεί πολύ ενδιαφέρον. Θέλουν όλοι οι συνάδελφοι να <clears throat> συμμετάσχουν. Δεν θέλουμε περισσότερα απόβλητα στις θάλασσές μας, δεν θέλουμε πιο πολλά απόβλητα από ψάρια και δυστυχώς προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έχετε το λόγο, κυρία Κόπιψκα, από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και όλους εσάς γιατί βλέπω ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους πολιτικούς στόχους αυτής της έκθεσης. Φαίνεται ότι έχουμε κοινούς στόχους, εσείς και εμείς, να σταματήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μόλυνση των θαλασσών. Ε, προτείνουμε ένα πακέτο μέτρων και σε σχέση με άλλα θέματα που αφορούν ε, μόλυνση από πλαστικά, παραδείγματος χάρη, και είναι ένα πρόβλημα παγκοσμίω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί αυτό που είπατε, ότι πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίσουμε τις πηγές της μόλυνσης, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται στην γη. Εδώ αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη μόλυνση που προκαλείται από τα πλοία. Και με την πρόταση αυτή θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να υπάρξει μια συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό ε, πλαίσιο κανονισμών και συμμόρφωση εκ μέρους όλων των κρατών μελών. Να υπάρξει πραγματική εφαρμογή, το είπατε κι εσείς. Θέλουμε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί μόνο έτσι θα τηρηθεί. Αναφερόμαστε λοιπόν σε διάφορες προτάσεις με την έμεση ε, επιβολή τελών και συμφωνώ μαζί σας ότι η πρόταση αυτή είναι αποτελεσματική. Είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ενθαρρύνουμε τα πλοία ουσιαστικά να τηρήσουν αυτό τον κανόνα, γιατί εδώ δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ της ποσότητας των αποβλήτων και του ποσού που πρέπει να καταβάλουν ε, τα πλοία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έτσι και αλλιώ αφού θα πληρώσουν, οι ποσότητες ε, τελικά θα ακολουθούν την καταβολή του ποσού προτείνατε κάποιες ε, προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι συμπληρωματικές. Συμπεριλαμβάνεται άλλου είδους απόβλητα όπως το έρμα, όπως τους, αυτά τα απόβλητα τα οποία ε, προορίζονται για τους scrubbers. Και βεβαίως ε, αυτές οι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να τηρηθούν. Παραδείγματος χάρη, τα υγρά τα οποία προέρχονται από τους scrubbers, πώς ακριβώς θα κατηγοριοποιηθούν στις κατηγορίες των αποβλήτων. Εμείς με μεγάλη χαρά θα συζητήσουμε περαιτέρω όλες αυτές τις υποκατηγορίες αποβλήτων και ποιες μπορούν να ενσωματωθούν. Επίσης άκουσα και κάποια άλλα σχόλια, κάποιες ερωτήσεις, προτάσεις όσον αφορά τους αποκλεισμούς. Παραδείγματο χάρη, τα μικρά λιμάνια. Σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας κατάλαβα ότι υπάρχει ενδιαφέρον να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Να μην υπόκεινται δηλαδή κάποια λιμάνια, τα μικρότερα, στην τήρηση αυτών των κανόνων. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στις προτάσεις ένα σχέδιο για την ε, διαχείριση των αποβλήτων με ένα πιο απλό τρόπο ενδεχομένως. Με όλο αυτό το... Ε, με όλες αυτές τις δυνατότητες, αν θέλετε, μπορούμε να υποχρεώσουμε τα λιμάνια να προβλέψουν ε, κάποιου ίδιους, ίσως απλούστερο τρόπο χειρισμού των αποβλήτων. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονό ότι κάποια λιμάνια ουσιαστικά έχουν μεγάλη κυκλοφορία αλλιευτικών σκαφών και θα πρέπει να δούμε αν συμπεριλάβουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ε, λιμανιών στα μικρά λιμάνια, αυτά δηλαδή που ε, εξαιρούνται από κάποιες από αυτές τις διατάξεις, από αυτούς τους κανονισμούς, θα δημιουργήσουμε ένα άλλο είδους πρόβλημα. Τώρα, με την ε, ναυτιλία μικρών διαδρομών, την ακτοπλοεία, short sea shipping, Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές ε, οι διαδρομές οι οποίες ουσιαστικά συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία για να μην αποκλειστούν πάλι ε, οι περισσότερες από αυτές τις διαδρομές από τις υποχρεώσεις για τα απόβλητα. Θα πρέπει λοιπόν πολύ προσεκτικά και εδώ να δούμε τι εννοούμε, να δούμε τους ε, ορισμούς. Το θέμα του απόπλου των πλοίων από το τελευταίο λιμάνι, πριν εγκαταλείψουν δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, απλώς θα πρέπει να σιγουρευτούμε 100% ε, να έχουμε δηλαδή απόλυτη εγγύηση ότι το λιμάνι προορισμού του πλοίου που εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ε, την διαχείριση των αποβλήτων. Υπάρχει επίσης και αναφορά στην ΕΜΣΑ. Πρόκειται για τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Εδώ σίγουρα θα χρειαστούν και κάποιες επιπλέον ε, νομοθετικές προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τις ε, απορρίψεις αποβλήτων στη θάλασσα, τις διαρροές, για να συμπληρωθεί και αυτό το νομοθετικό κείμενο. Κοιτάω λίγο και το χρόνο που έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Δεν ξέρω. Ε, ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις. Αν κάτι ξέχασα, με μεγάλη χαρά θα σας απαντήσω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον στην Επιτροπή και βεβαίως θα επεξεργαστούμε το κείμενο και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να πω ότι ε, ε, ε στον συνάδελφο ότι πραγματικά είναι σημαντικό το ότι ανέφερε σε, ε, τη Μαρπόλ, είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τη Μαρία. Ε, ναι, δεν είναι τώρα πια στην αλλά πράγματι έχει δίκιο ε, το να δούμε πόσο μπορεί να γίνεται αυτή η συμπερίληψη και των πλωτών εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιμήκυνση των σχετικών ε, ε, προθεσμιών, να πω από τώρα ότι δεν συμφωνώ, γιατί όσο πιο γρήγορα επιτύχουμε το νέο σύστημα, τόσο το καλύτερο. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο Πίτερ, σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα συλλογή των αποβλήτων στου ποταμού, θα μπορούσε να μα πει λίγο παραπάνω το τι ήδη δηλαδή κάνουν τα κράτη προκειμένου να το επιτυχάουν από σήμερα. Πάντω, ευχαριστώ για την επιβεβαίωση των όσων έδωσε σε σχέση με αυτά που κάνω. Και τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, ε, πλατφόρμες αυτές που ανέφερες και τη συμπερίληψή τους, ναι, ε, αυτές οι πλατφόρμες offshore κατά κάποιο τρόπο θεωρούνται ως πλοία, αλλά το ζήτημα εδώ είναι τα απόβλητα των πλοίων και όχι των πλατφορμών offshore. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, ο ΕΜΣ αναφέρθηκε ήδη. Μετά, συνάδελφος από την ΚΟΕ, δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα, στο συγγνώμη, πάντως σε ό,τι αφορά τους ορισμούς πράγματι θα πρέπει ε, να δούμε ακριβώς και να ορίσουμε το τι είναι για παράδειγμα ένας μικρός ε, απόμακρος λιμένα ή τι είναι μικρών αποστάσεων αυσυπλοεία και ε, οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ξέρουμε από την Επιτροπή Αλληλεία ότι η τι είναι μικρών αποστάσεων, ναυσιπλοεία και οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ξέρουμε από την Επιτροπή Αλία ότι η Europes έχει υποβάλει μια σειρά από προτάσει τροπολογιών που θα μπορούσαν να γίνουν, οπότε θα ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, ξέρουμε ότι και από την Επιτροπή Αλία θα υπάρξουν τροπολογίε που θα υποβληθούν. Από εκεί και μετά θα πρέπει πράγματι να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα στα ενεργά και τα παθητικά αλλιευόμενα ε, απορρίμματα, ε, απόβλητα και πράγματι θα πρέπει να λάβουμε επίση υπόψη μα και τι συνέργειε, ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ικανοτήτων που έχουμε. Και αυτό είπε και εμένα, δηλαδή ότι ε, δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται υπερβολικά οι μικροί λιμένε και θα πρέπει να συνεργάζονται, για παράδειγμα, μεγαλύτερες ε, λιμένες. Ε, πράγματι θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μία αποτελεσματική λύση εδώ, λαμβάνοντα υπόψη και τι διαφορετικέ μα απόψει. Τώρα, ε, ό,τι αφορά το ζήτημα των τιμών, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ, ω Επιτροπή, μπορεί να σου απαντήσει. Νομίζω πω οι τιμέ καθορίζονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αλλά δυστυχώ αυτό είναι το μόνο που ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Πάντω, ε, σε ό,τι αφορά τα σχόλια που έκανε η Επιτροπή, το θεωρώ θετικό και ήδη το συζητήσαμε, ότι ε, παρότι ε, συμφωνούμε σε γενικέ γραμμέ με την πρόταση τη Επιτροπή. Έχουμε και κάποιε τοπολογίε. Πραγματικά είναι θετικό αυτό και θα τι υποβάλουμε. Πάντω, σα ευχαριστώ όλου εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση και είμαι πεπισμένο ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκέζινε Μάισνερ. Προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών 18 Ιουλίου το μεσημέρι στις 12. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στη δημόσια ακρόασή μας. Οι διακρίσεις στον διάβλο διανομής αερομεταφορέων. Θα παρακαλέσω τους προσκεκλημένους μας να έρθουν στο Προεδρείο. Κύριε Ντεμπλέστ, κύριε Πάγκο και κύριε Νόλαν. Κύριε Άουρφ, ελάτε δίπλα μου.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 Συνάδελφοί μου, τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα ουσιώδου σημασία για το μέλλον των μεταφορών συγκεκριμένα της αεροπλοείας και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα διάφορα δίκτυα διανομής υπηρεσιών στις αερομεταφορές. Το θέμα αυτό άπτεται πολλών διαφορετικών πτυχών, όπως η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια, η μη ε, ε διάκριση στις τιμές, Κάτι που μας έρχεται πολύ εύκολα στο νου, ιδίως επειδή έχουμε συχνά τη συζήτηση της θέσπισης ε, πλέον τέλους ε, πώληση από διάφορου αερομεταφορεί αφού το επιπλέον τέλο, όταν η πώληση του εισιτηρίου δεν περνάει από το δικό του στο ηλεκτρονικό σύστημα. Με τη χάρτα λοιπόν ε, και τον κωδικό καλή συμπεριφορά ΣΕΡΕΣ, θα πρέπει όλα αυτά κάπως να αντιμετωπιστούν. Θα θέλαμε λοιπόν με την ακρόαση αυτή να έχουμε μια πανοραμική εικόνα της σημερινής κατάστασης του όλου αυτού κλάδου, της διανομής και της παροχής αεροπορικών υπηρεσιών, αερομεταφορών συγκεκριμένα. Είμαστε ε, ε, και διανύουμε μια πραγματική επανάσταση διότι αλλάζει τόσο η συμπεριφορά των καταναλωτών όσο και υιοθετούνται νέε τεχνολογίε. Το να κλείσει κανεί ένα εισιτήριο ή μια ε, υπηρεσία αερομεταφορέα, όπω λέγεται, είναι μια εμπειρία τελείω διαφορετική πλέον από την πλή αγοραπολισία που γνωρίζαμε πριν από κάποια χρόνια. Είναι πολλέ εταιρείε, διαφορετικά τα συστήματα που χρησιμοποιούνται και διαφορετικά τα είδη υπηρεσιών. Είναι πιο πολύ άριθμα, πιο αποτελεσματικά, πιο εύκολα να τα έχει κανεί και φθηνότερα, Πιο ε, φορητά, πιο προσωποποιημένα, αλλά και πιο. Ε, ε, ε, περίεργα για τα προσωπικά μας δεδομένα. Εδώ λοιπόν με αυτές τις ε, μεταβολές και αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πλέον εκτήματα συνοδεύονται και από πολλούς κινδύνους. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν με αυτήν την μεγάλη ομάδα πυρογνωμόνων να καλύψουμε μια σειρά από συναρπαστικά θέματα. Και γι' αυτό στο πρώτο μας ε, γύρο θα ασχοληθούμε με το LN Distribution Channel, A Brief History. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Hours, ο οποίος είναι επικεφαλής των ε, νέων, ε, του νέου διάβλου διανομής. Είστε μέλος της ΙΑΤΑ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κύριε Ντεμπλούστ, είστε Γενικός Γραμματέας και εσείς και εκπροσωπείτε την Ένωση Ευρωπαίων ε, Ταξιδιτικών Πρακτόρων και ε, Tour Operator. Μετά έχουμε τον κύριο Στεφάν Παγκό, ο οποίος είναι και αυτός Γενικός Διευθυντής και συνειδητής της Flying. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Και μετά ο κύριος Μάρτιν Νόλαν, ο οποίος ε, είναι Διευθυντής της Sky Scanner στο Τμήμα Νομικών και Εταιρικών Υπηρεσιών και ανάπτυξή τους. Καλώς ήρθατε να διοργανώσουμε κάπως τη συζήτηση, διότι έχουμε περιορισμένο χρόνο. Θα ζητήσω τον καθέναν ομιλητή να μας ε, κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Έχετε 7 λεπτά ο καθένας και εγώ θα ελέγχω το ρολόι. Δεν θα κάνω δωράκια. Θα είμαι το ίδιο αυστηρή και με τους βουλευτές και με το δεύτερο γύρο και τη στρογγυλή, το δεύτερο πάνελ. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Εμπρός. Good afternoon, Olivier. I'm working for IATA, International Air Transport Association. Ναι, ε, ε, εκπροσωπώ την, ε, την Ένωση των Αερομεταφορών και εκπροσωπούμε εδώ μία σειρά από επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπούν ένα σημαντικό ποσοστό των αερομεταφορών. Serious activities. Next slide. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την διανομή και ένα θέμα μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών και των καταναλωτών. Ε, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες πρακτορείων. Ε, οι αεροπορικές εταιρείες ε, και το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τα πρακτορεία, για τις κρατήσεις των πτήσεων και τον καθορισμό των τιμών. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, τρία CRS σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Amadeus με 65% κάλυψη. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, το CRS καλύπτει 80% των Και πολλές φορές υπάρχει μία και μοναδική ε, τέτοια χρήση αυτών των ε, συστημάτων. Πολύ σπάνια υπάρχει διαφορετική χρήση των CRS. Και διαπιστώνουμε ότι εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, δολάρια ουσιαστικά περνάνε <clears throat> μέσα από τα συστήματα κρατήσεων αυτά. εκατομμύρια αν θέλετε να δούμε παγκοσμίω. Οι διάφοροι πράκτορες βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα και μπορούν πολύ εύκολα να περάσουν από το ένα στο άλλο η κάλυψη αυτών των αναγκών στοιχίζει περίπου 40 ευρώ για, ένα, για μια πτήση ε, αλέρετουρ και επιπλέον οι συμβάσεις αυτές, οι οποίες ονομάζονται πλήρες συμβάσεις ε, για το σύστημα αυτοκρατήσεων, επιτρέπουν να γίνονται πολλές συναλλαγές βάσει των συμβάσεων αυτών και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κανάλια, ε, ιστοσελίδες ε, και άλλες δυνατότητες που ε, παρέχει το διαδίκτυο. Είναι σχεδόν αδύνατον για μια αεροπορική εταιρεία να διαπραγματευτεί με ένα σύστημα CRS, καθότι το κόστος και οι όροι ουσιαστικά μονομερώς επιβάλλονται. Βλέπουμε επίσης ότι το ίδιο κάνουν και τα πρακτενία. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση η κάθε αεροπορική εταιρεία ουσιαστικά να ε, έχει σύμβαση με όλα τα συστήματα CRS. Τώρα, ποια είναι τα συστήματα αυτά που επιτρέπουν στον, τελευταίο καταναλωτή, στον τελικό συγγνώμη, καταναλωτή να έχουν ε, πλήρη γνώση ε, αυτού που συμβαίνει. Εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουν ε, αναπτυχθεί εναλλακτικές τεχνολογίες όπως ε, το σύστημα New Distribution Capability, ένα νέο σύστημα για τη χωρητικότητα, το NDC, το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή να έχει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβασή του σε νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και βλέπουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δαπανίσει δισεκατομμύρια σε αυτές τις νέες δυνατότητες και τεχνολογίες, δεν μπορούν όμως να τα χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν. Βλέπουμε επίσης ότι τα συστήματα CRS μέχρι του χρόνου θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες. Τα CRS όμως συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ίδιες εμπορικές πρακτικές. Και αν θέλουν οι αεροπορικές εταιρείες να ξεφορτωθούν ουσιαστικά αυτές τους περιοριστικές ε, ρήτρε, δεν έχουν σήμερα απολύτως καμία άλλη επιλογή από το να υπομισθούν το επιπλέον κόστος εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο σήμερα CRS. Είναι το λεγόμενο, αν θέλετε, κόστος CRS. Γι' αυτό και μέσω διαφορετικών δικτύων ε, προσπαθούν να βρουν τα πρακτορία διαφορεστικές ουσιαστικές εναλλακτικέ λύσεις με χαμηλότερο κόστος. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν όμως τέτοιες επιλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικός ανταγωνισμός. Τα CRS θα πρέπει να ξεκινήσουν συναλλαγές σε χαμηλότερο κόστος, κάτι το οποίο θα επιτρέψει περισσότερες δυνατότητες. Η ΙΑΤΑ πιστεύει ότι αυτό θα είναι πολύ καλό για τον καταναλωτή, ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός, περισσότερη διαφάνεια, ουσιαστικά θα επιτρέψουν καλύτερη και οικονομικότερη πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι καταναλωτές, οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ίδιες τιμές μέσω διαφορετικών ε, δικτύων. Και θα πρέπει να πάρουν την απόφαση μέχρι να τελειοποιηθούν και να ολοκληρωθούν τα συστήματα CRS να μπορούν να χρησιμοποιούν μια εναλλακτική τεχνολογία. Υπάρχει σήμερα μεγάλη δυσαρέσκεια από μέρους των αεροπορικών εταιριών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις καθυστερήσεις για την ε, ενημέρωση των συστημάτων CRS. Σήμερα είμαστε σε έναν ανταγωνισμό ο οποίος ε, είναι στρεβλωμένος και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες στον καταναλωτή. Υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση, η οποία σε καμία περίπτωση όμως δεν οφείλεται στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά στα συστήματα CRS. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Άουρς. Πραγματικά σεβαστήκατε και το χρόνο ομιλία σα. Συγχαρητήρια. Και τώρα εσεί, κύριε Ντεμπούστ. Thank you, Madam Good afternoon. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Εκπροσωπούμε τους 70.000 ε, online ταξιδιωτικούς πράκτορες, φυσικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλους tour operators οι οποίοι παρέχουν ε, ταξιδιωτικές υπηρεσίες ε, αξίας, για παράδειγμα πέρσι, μόνο ε, ύψους 210 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Καταρχήν, πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια η παροχή των υπηρεσιών και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες προβαίνουν σε marketing όχι μόνο αεροπορικών εταιριών, αλλά και άλλων επιχειρήσεων, για παράδειγμα ξενοδοχείων, ε, μίσθωση αυτοκινήτων, ε, σε δρόμο και ούτω καθεξής. Και βέβαια, κατά τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί μια νέα διάσταση, καθώς έχει προσθεθεί ένας νέος διάβλος ε, πώληση και φυσικά, δηλαδή online και φυσικά οι Ευρωπαίοι καταναλωτές προτιμούν αυτήν την ε, προσέγγιση αν θέλετε της νέας δηλαδή της ε, εξυπηρέτησής τους ε, μέσω ενός κοινού παρόχου υπηρεσιών. Τώρα, περνάμε εδώ στους σιδηροδρόμους. Εδώ Έχουμε για παράδειγμα το σύστημα των, το αεροπορικό όπου έχουμε τα συστήματα τα οποία ενοποιούν ε, την διαχείριση, πράγμα το οποίο έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Καταρχήν, με αυτόν τον τρόπο οι αεροπορικές εταιρείε έχουν ένα ενιαίο σύστημα το οποίο ε, ε, επιτρέπει στα 70.000 μέλη να έχουν πρόσβαση στο GTS και κατά συνέπεια να έχουν πρόσβαση στους καταναλωτές προσφέροντάς τους πολύ προσιτές τιμές. Άρα λοιπόν τα GTS αποτελούν ουσιαστικά ένα τρόπο πρόσβαση ε, σε αυτόν τον ε, ε, διάβλο διάθεση των προϊόντων παρέχοντας τη σύγκριση των τιμών αλλά και διάφορε λειτουργίες κράτηση και πώληση εισιτηρίων. Και ενώ παρέχεται η δυνατότητα αμερόληπτης και ανεξάρτητης σύγκριση των τιμών. Και βέβαια ε, το, εκείνος που υποφελούνται κυρίως από αυτήν την αλυσίδα αξίας αν θέλετε είναι ο καταναλωτές αφού έχει πλήρη και συνοπτική εικόνα της κατάστασης των τιμών. Ωστόσο η κατάσταση έχει καταστεί λίγο πιο περίπλοκη κατά τελευταία χρόνια. Οι βετεράνοι λοιπόν ε, σε αυτό το τομέα θυμόμαστε τους παλιούς καλούς καιρούς όπου αγοράζαμε ένα εισιτήριο και αναμέναμε ένα γεύμα, ένα ποτήρι κρασί ε, μία αποσκευή 20 κιλών και όλα αυτά να περιλαμβάνονται μέσα στη τιμή του εισιτηρίου. Σήμερα με αυτό το unbundling όπως λέγεται αυτών των εισιτηρίων, των αεροπορικών ειδικότερα, θα πρέπει κανείς να πληρώσει ξεχωριστά το εισιτήριο, από εκεί και μετά να πληρώσει την αποσκευή του, να πληρώσει το κάθισμά του και ίσως ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, πληρώνουμε και ένα τέλος για την ύπαρξη πιλότου πάνω στο αεροσκάφος. Όλα αυτά υποτίθεται πως συμβάλλουν στην βελτίωση της εμπειρίας ε, του καταναλωτή, του επιβάτη, αλλά νομίζουμε πως εδώ πρόκειται για μια ζούγκλα τιμών, τελών και ε, φόρων. Οπότε στο πλαίσιο ε, ειδικότερα ε, το ΦΠΑ θεωρούμε πως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις τιμές που υπηρετούν στην αγορά. Και εδώ περνάω στην επόμενη διαφάρα και στο NDC. Τι θα λέγατε για την ιδέα να μπαίνετε στο αγαπημένο σας σούπερ μάρκετ, να κάνετε ε, να, να, να κάνετε ένα swipe ε, μια κάρτα όπως μπαίνετε ε, και να σας δείχνει αυτόματα τις επιτροπέ που επιθυμεί το σούπερ μάρκετ. Αυτό ακριβώς είναι το σκεπτικό για παράδειγμα που εφαρμόζεται ήδη από την Amazon και το οποίο είναι το NDC. Δηλαδή συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα στο πλαίσιο του NDC προτού καταδειχτεί η, η, η τιμή Ενό εισιτηρίου. Αυτό δημιουργεί βέβαια ζητήματα σε ό,τι αφορά την ε, διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα των τιμών, το ζήτημα τη διαχείριση των δεδομένων και αυτό ειδικότερα όταν αυτά τα δεδομένα ε, δεν ε, κατευθύνονται και δεν αφορούν μόνο τις συγκεκριμένου αερομεταφορεί, αλλά και άλλους. Και ευτυχώς τα περισσότερα GTS μετατρέπονται πλέον σε έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα νέα πρότυπα. Πάντως υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο του νέου συστήματος. Ε, ποιο είναι λοιπόν το διακύβευμα εδώ, ποιες είναι οι τέσσερις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο μιας μελλοντική αναθεώρησης ε, δύο σημαντικών κανονισμών, δηλαδή του κανονισμού 208 σε ό,τι αφορά τις εναέρες μεταφορές ε, και μετά τον 80 ε, του 2019 ε, σε ό,τι αφορά την ε, διοντολογία σε αυτόν τον τομέα. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή προετοιμάζει την αναθεώρηση αυτών των δύο κανονισμών για του χρόνου. Και οι τέσσερι προκλήσει λοιπόν τι οποίε θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο νομοθέτη είναι εξή. Καταρχήν, η διατήρηση τη πλήρου πρόσβαση στι τιμέ. Ακούσαμε από τον κύριο Άουερ το γεγονό ότι δεν επιθυμούν οι αερομεταφορεί την πλήρη ε, πρόσβαση στις τιμές τους γιατί δεν τους αρέσει οι επιβάτες να μπορούν να κάνουν ε, σύγκριση των τιμών. Από εκεί και μετά θα πρέπει να διατηρηθεί η διαφάνεια ε, των τιμών των εισιτηρίων και κατά συνέπεια της συγκρισμότητας των τιμών των εισιτηρίων. τρίτον, θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τον διάβλο που θα επιλέξει. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει είτε από τον αερομεταφορέα είτε μέσω έμεσου διάβλου. Διάθεση των εισιτηρίων. Και μια τέταρτη πολύ σημαντική πρόκληση είναι το να αποφευχθεί η διάκριση των καταναλωτών με βάση, για παράδειγμα, το κράτος μέλος της κατοικίας τους, αλλά ε, και με βάση ε, το κράτος μέλος της έδρας ε, του διανομέα των εισιτηρίων. Αυτά λοιπόν, αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά αν θέλουμε να επιτύχουμε τη διατήρηση του κοινού ευρωπαϊκού ουρανού, του Single European Sky. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά συμπεράσματα και μηνύματα που θέλω να περάσω στη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχετε εσείς, κύριε Στεφάν Πενγκό. Και εσείς για 7 λεπτά. Είστε έτοιμο, πάμε. Εκτός μικροφώνου κύριο Πενγκό. Καλησπέρα σα. Σα σας ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα. Είμαι συνειδητής και γενικός διευθυντής της ε, Flying ε, που έχει έδρα στο Βερολίνο και δίνει στους λιανοπολιτές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν προϊόντα για την κράτηση εισιτηρίων μοναδικά και ε, εύκολο να διασυνδεθούν στις προσωπικές ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Βλέπετε στην οθόνη το μοντέλο της πώληση εισιτηρίων τα τελευταία 30 χρόνια. Το μοντέλο αυτό το ονομάζω αυτό που βασίζεται στους ε, διαμεσολαβητές. Δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα ε, Σέρπα, Travelport, ε, Amadeus και οι πελάτες τους, Expedia, Opondo και άλλες εταιρείε που πολλούν. Αυτοί που ασχολούνται με όλες τις συναλλαγές μεταξύ των οποίων και οι πληρωμές. Βάσει του περιεχομένου που έχουν φορτωθεί στην βάση δεδομένων των ΗΠΑ λόγω χάρη ATP και των ATP ε, μάλλον και των ε, χρονοθυρίδων των πραγμάτων. Πώς δουλεύει αυτό, ας πούμε, ότι είσαστε στις Βρυξέλλες και θέλετε να πάτε στη Νέα Υόρκη. Πάτε στο Expedia. Βάζετε τις παραμέτρους σας, ε, ημερομηνίες, διαδρομολόγιο, πόσοι επιβάτες και κάνετε την αναζήτησή σας. Τι συμβαίνει εκεί, το GTS αναζητά τους ναύλους από το EG και το ATPCO και το μόνο που κάνουν με την αεροπορική εταιρεία είναι να ρωτήσουν αν η νάυλη είναι ακόμα διαθέσιμοι. Την ε, προσφορά λοιπόν την κάνει η GDS. Η αεροπορική εταιρεία δεν γνωρίζει ότι ψάχνεται. Πρώτο σημαντικό. Μόλις ε, κλικάρει κανείς στο κράτηση, τότε το GDS δημιουργεί την κράτηση στο δικό του σύστημα, εκδίδει το εισιτήριο και η Expedia παίρνει τα χρήματα χρεώνοντας την πιστοτική. Αυτό είναι το σημερινό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί καταπληκτικά με του συγκεκριμένου πληρωτέ, του operator, τα ταχυδρομικά πρακτορία, του Consolidator, όπω ονομάζονται. Όμω για τον πελάτη είναι άγνωστη η περιπλοκότητα του όλου συστήματο. Το μοντέλο λοιπόν αυτό που είδατε λειτουργεί πολύ καλά όταν οι αεροπορικέ ε, εταιρείε μπορούσαν να διαπραγματευτούν και να εμπορευτούν το προϊόν τους. Όμως έναν κόσμο όπου ο καθένα εμπορεύεται το προϊόν του περισσότερο προϊόν και όχι ω μια δυνατότητα, μια υπηρεσία, τότε περιορίζεται το σύστημα αυτό έχει όρια. Για παράδειγμα, οι εταιρείε, οι αεροπορικέ εταιρείε δεν μπορούν να ελέγξουν την προσφορά που βλέπετε εσεί στο Expedia. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει πελάτη που ψάχνει. Ε, μπορούν να στείλουν για πώληση κάποια από τα προϊόντα του, αλλά δεν μπορούν να προσφέρουν όλε τι υπηρεσίε που θέλουν. Επίση, δεν μπορούν να αποστασιοποιηθούν ή μάλλον να διαφοροποιηθούν από τι ανταγωνιστικέ εταιρείε. Δεν έχουν τα στοιχεία. Ε, η συνέπεια όλων αυτών των περιορισμών ε, επηρεάζει τον τελικό καταναλωτή. Εάν είστε καταναλωτή που ψάχνει στο Expedia, είναι αδύνατο να πάρετε το πλήρες κόστο τη εταιρεία σα μαζί με τι υπηρεσίε που μπορεί να είναι σημαντικέ για εσά. Α πούμε το έγκαιρο check-in, η επιλογή θέση. ή ένας ναύλος που είναι σχετικά ευέλικτο γιατί δεν ξέρετε σίγουρα τι ημερομηνίε σα. Είναι αδύνατο να έχετε πλήρες, πλήρη εικόνα του κόστους πριν κάνετε την κράτηση. Έπειτα, ε, ας πούμε ότι αν θέλετε να τα κρατήσετε ε, για ένα διάστημα, δεν γίνεται. Ο ναύλος είναι διαθέσιμος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ε, σκεφτείτε τι γίνεται όταν ε, πολλούνται ναύλοι 500 ευρώ και τη συγκρίνετε με κάτι άλλο. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή. Επίση, τι περιλαμβάνεται, μία αποσκευή, δύο αποσκευέ, τι θέση μπορεί να παρει κανει κανείς, Wi-Fi έχει το αεροσκάφο και το καθεξής. Αυτά δεν τα ξέρει όταν αγοράζει. Και επίσης, όταν αγοράζει κανεί δεν ξέρει από πού αγοράζει, από ενδιάμεσο, από αεροπορική εταιρεία, δεν υπάρχουν διευκρινήσει. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ λοιπόν στη Flying δημιουργούμε ένα νέο σύστημα διανομή επιρροσίων μεταφορών, ε, όπου πηγαίνουμε στου μεταπράτε ε, και προσπαθούμε με έναν απλό τρόπο να πουλήσουμε εισιτήρια στον τελικό χρήστη απευθεία, χωρί να περνάμε από το περίπλοκο, ε, την περίπλοκη εργάνωση του σημερινού σύστηματο. Αυτή η νέα πλατφόρμα βασίζεται σε ένα μοντέλο που κέντρο έχουν την αεροπορική εταιρεία και την ευθύνη την αναλαμβάνουν οι εταιρείε, την αναζήτηση, την ε, κράτηση, ε, τι πληρωμέ, την κράτηση θέσεων. Εάν λοιπόν κλικάρει κανεί Βρυξέλλε-Νέα Υόρκη, στην αναζήτηση αμέσω, στέλνονται μηνύματα απευθεία ή αμέσω ε, στι αεροπορικέ εταιρείε. Αυτέ συγκεντρώνουν όλε τι πληροφορίε, βλέπουν όλε του ναύλου και κάνουν τι προτάσει του. Όταν λοιπόν στη δική μα πλατφόρμα κάνει αυτό κανεί κανείς αυτή την αναζήτηση, βλέπει όλου του διαθέσιμου ναύλου. Διαλέγει τον ναύλο που του αρέσει καλύτερα, επιλέγει την αεροπορική εταιρεία που δίνει αυτόν τον ναύλο, κλείνει το εισιτήριο και ε, έτσι χρεώνεται η κάρτα του. Το μοντέλο αυτό ε, πηγαίνει πολύ καλά με τους ε, όπω λέω εγώ, παράγοντες. Ε, δείτε το Facebook ή το TripAdvisor. Όποια εταιρεία πλατφόρμα θα θέλει να δημιουργήσει τη δική της εσωτερική, ε, το δικό της εσωτερικό εργαλείο κρατήσεων. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή που να πουλήσουν ε, πτήσεις, γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Πιστεύουμε ότι το μοντέλο αυτό θα γίνει ο κανόνας και ο καθιερωμένος πληρωτής, όπως μπορούμε να το πούμε, θα είναι το κέντρο όλων των αγοραπολισιών. Ε, σκεφτείτε τι γίνεται με αυτό το μοντέλο, εάν μεθαύριο το TripAdvisor και το Facebook αρχίσουν να πουλούν πτήσει. Το δίκτυό του θα είναι πολύ μεγαλύτερο από όλου του προηγούμενου. Θα έχουν περισσότερο εισόδημα και το εισόδημα αυτό θα πηγαίνει απευθεία από τι πωλήσει και θα μπορούν να ε, το πάρουν κατευθείαν οι αεροπορικέ εταιρείε. Ε, για του μεταπράτε, θα είναι πολύ εύκολο να οργανώσουν ένα σύστημα ε, πτήση κράτηση. Διότι τώρα για να, για να πάρει έγκριση κάποιο ταξιδιωτικό πράκτορα δεν είναι απλό. Ε, παίρνω ε, τηλεφωνήματα από νεοφυεί εταιρείε συνεχώ που μου λένε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα σα για να πουλήσουμε εισιτήρια γιατί δεν έχουμε έγκριση. Για τον τελικό καταναλωτή θα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί πραγματικά μπορεί με μία σελίδα να δει όλου του ναύλου και να του εγκρίνει. Θα σα ήθελα να σα δείξω τη σελίδα για να το καταλάβετε. Ο καταναλωτή καταλαβαίνει τι αγοράζει όταν αγοράζει. Μπορεί εύκολα να συγκρίνει μεταξύ των διαφορετικών προσφορών των διαφορετικών εταιριών, ακόμη και αν οι εταιρείε εμπορεύονται τα προϊόντα με διαφορετικό τρόπο. Και τελικά μπορεί να κάνει μια ε, ε, απόφαση βάσει στοιχείων. Να πάρει μια απόφαση βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι επενδυτέ δεν θέλουν να μπουν στη διανομή υπηρεσιών αερομεταφορών. Ψάχνουμε τρία χρόνια. Έχουμε στο Διοικητικό μα Συμβούλιο προσκαλέσει μέχρι και γενικού διευθυντέ αεροπορικών εταιριών. Κανεί δεν θέλει να δώσει χρήμα για το δικό μα δίκτυο. Οι μόνοι που θέλουν είναι τα hedge funds τη Νέα Υόρκη που θέλουν να ρισκάρουν τα λεφτά του. Γιατί? Γιατί ε, είναι εύκολο να βάλει κανεί να θέσει στην αγορά μια τέτοια πλατφόρμα. Οι περισσότεροι επενδυτές, η πλειοψηφία των ε, ε, επενδυτών βλέπουν το GDS ε, ως μια πολύ ισχυρή ομάδα με ατελείωτη εξουσία. Εδώ πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό. Διότι εάν σκεφτούμε το Booking.com, το Expedia και όλα τα σχετικά, το eDreams, το Opondo, είναι τρόποι να πάρει κανείς στα χέρια του να σφετριστεί τον πλούτο και όχι να, ε, πάρει, να αφήσει να φύγουν πελάτες αλλού. Ευχαριστούμε κύριε Παγκό. Δεν είδαμε ότι πέρασε ο χρόνος γιατί ήσασταν ε, συνεργαστικός. Κύριε Νόλαν, παρακαλούμε για να ολοκληρώσουμε αυτό το πάνελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που καλέσετε και την Sky Scanner μπορώ και εγώ να συμμετάσχω. Πολύ σύντομα, ποιοι είμαστε. Είμαστε μια πλατφόρμα έρευνας, 17, 70 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτονται την πλατφόρμα μας και φυσικά 1200 ε, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες συμμετέχουν με 2.003 ε, χρόνο ίδρυσης και 1.100 άτομα που εργάζονται στην πλατφόρμα μας παντού στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι το Sky Scanner είναι ένα σύστημα σύγκρισης και ε, εξέβρεσης της καλύτερης τιμής. Καταρχήν, ποια είναι η πρώτη, αν θέλετε, θετική συνέπεια αυτού του συστήματος. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον να συγκρίνει. Ένας καταναλωτής που με διαφάνεια γνωρίζει, είναι ενημερωμένος, μπορεί να κάνει την καλύτερη επιλογή. Είμαστε, αν θέλετε, συνδεδεμένοι με πολλές αεροπορικές εταιρείες, με πολλούς φορείς παροχής υπηρεσιών και μπορούμε να διαπιστώσουμε ακριβώς ποιες είναι οι τιμές προσύγκριση και να δώσουμε τις περισσότερες πληροφορίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο καταναλωτής, ο χρήσης των υπηρεσιών μας να μπορεί να κάνει την καλύτερη επιλογή έχοντας τις περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό και του παρέχουμε ε, κάθε είδους πληροφορίες και βεβαίως παρέχουμε στην ιστοσελίδα μας και τη δυνατότητα για διαφήμιση. Οι συνάδελφοι στη σημερινή συζήτηση ε, παρουσίασαν κάποια από τα στοιχεία που μας αφορούν, τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες, ε, διανομής, η τεχνολογία η οποία βεβαίως έχει οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή στα συστήματα διανομής ε, τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τεχνολογίας και σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις διαπιστώνουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες κερδίζουν μερίδιο της αγοράς στα δίκτυα διανομής. Υπάρχει ανταγωνισμός βεβαίως και παρακολουθήσατε τον ανταγωνισμό αυτό όχι μόνο από τις εταιρείες χαμηλού κόστους, low cost αεροπορικές εταιρείες, αλλά από την άλλη μεριά ο καταναλωτής σήμερα βρίσκεται σε μια σύγχυση όταν ε, δεν ξέρει ακριβώς τι προϊόντα συγκρίνονται, αν πρόκειται δηλαδή για όμοια προϊόντα, συγκρίσιμα προϊόντα. Εμείς ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε, επαναλαμβάνω στον καταναλωτή, ότι δεν υπάρχει παραπληροφόρηση και ότι πραγματικά η σύγκριση γίνεται μεταξύ συγκρίσιμων προϊόντων. Όσον αφορά την καινοτομία και την τεχνολογία, ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Όταν κάποιος ε, θέλει να ενημερώνει τον καταναλωτή και να τον ενημερώνει έτσι ώστε να μπορέσει να κατανοήσει καλύτερα ποιες είναι οι αναλλακτικέ λύσεις τις οποίες καλείται να επιλέξει. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώσουμε τον ε, ταξιδιώτη, τον επιβάτη, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι συγκρίνουν ε, ε, σε αυτή την ε, μεταέρευνά τους διαφορετικές πλατφόρμες, διαφορετικά στοιχεία και αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό πέρα από την έρευνα, την κράτηση είναι και το θέμα των πληρωμών, ο απόρριτος χαρακτήρας των δεδομένων των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα για κάποιες από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακές τεχνικές. Υπάρχουν βεβαίως και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές τεχνολογίες και να μην στραφούν προς τον ψηφιακό κόσμο. Αυτό που ιδιαίτερα σήμερα εξετάζουμε είναι τις κανονιστικές διατάξεις, την ομοθεσία που διέπει αυτές τις πλατφόρμες. Επαναλαμβάνω ότι σκοπός μας είναι η καλύτερη ενημέρωση και η διαφάνεια για τον καταναλωτή. Σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ε, εμπλεκόμενων μερών, όπως σας εξήγησα, πρόκειται για μια αγορά η οποία πραγματικά σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τη τεχνολογία. Η εταιρεία Sky Scanner ουσιαστικά παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου. Ο σκοπός μας όμως είναι να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, να κατανοήσει ο καταναλωτής, ο πελάτης, με ποιο τρόπο μπορεί πραγματικά να επιλέξει την καλύτερη για αυτόν λύση, πού οφείλεται το κόστος και βεβαίως υπάρχει και μια πάρα πολύ σημαντική ενημέρωση από μέρους του καταναλωτή όσον αφορά την εμπειρία του. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τα σχόλια των ε, χρηστών. Το θέμα του χρήστη, του καταναλωτή καθοριστικό στοιχείο για μας, όπως σας είπα ήδη, είναι η διαφάνεια. Ότι δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι, ότι δεν υπάρχουν ε, ποσά τα οποία ουσιαστικά καταβάλλονται σε ενδιάμεσους και ότι το κόστος είναι κατανεμημένο ακριβώς όπως το παρουσιάζουμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες, της εναλλακτικέ λύσεις, να κατανοεί τις πληροφορίες που του δίνουμε για να μπορεί να κάνει την καλύτερη για αυτόν επιλογή. Θέλουμε λοιπόν να δίνουμε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα περιεχόμενα, σε όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Ε, με σκοπό να διασφαλίσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νόλαν. Σας ευχαριστούμε και για όσα μας είπατε. Να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε Κάμπ, κύριε Κλούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τι ομιλίε σα. Είναι πολλέ οι πληροφορίε αυτέ που θα πρέπει να κάτσουμε να τι μελετήσουμε για να τι αφομοιώσουμε. Πάντω, από δική μου πλευρά και για πολλού συναδέλφου, φαντάζομαι, η, το ανοιχτό πνεύμα και η διαφάνεια για τον καταναλωτή είναι ισόδου σημασία. Γιατί πολλοί από εμά απευθεία του καταναλωτέ, του πολίτε, να εκπροσωπούμε. Αυτό μα απασχολεί λοιπόν. Η αεροπλοεία στην Ευρώπη μας κάνει περήφανους και έχει ωφελήσει τους καταναλωτές. Η Ευρώπη ήταν ε, καλή σε αυτό. Κατάφερε να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός και ένομο, εντός νόμου. Ε, νομίζω ότι όλοι έχουμε βέβαια μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά κοινό στόχο. Μερικές παρατηρήσεις για την τελευταία ομιλία. Ή θα, απαντήσετε στο τέλ, θα απαντηθούν στο τέλος οι ερωτήσεις, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κάντε τις παρατηρήσεις σας και μαζί θέστε και τις ερωτήσεις σας. Να μας πείτε παρακαλώ κύριε Ούρς, γιατί λέτε ότι δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός στη διανομή. Ε, υπάρχουν μόνο τρεις ε, Και αναφέρατε και τον όρο συμφόρηση ε, στην αρχή της ε, ομιλίας σας. Ε, με συγχωρείτε και ωραίες κύριε Ντεμπούστ. Ε, μιλήσατε για τις κατήσεις και τους περισσότερους ε, ταξιδιωτικούς πράκτορες. Στην ουσία θέλετε περισσότεροι ουσιαρές να υπάρχουν σε ανταγωνισμό με όλα αυτά τα στρώματα που υπάρχουν μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του καταναλωτή στην ουσία για την παροχή των υπηρεσιών. Και τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει διότι είπαν ότι δεν θα ασχοληθούν με την προσφυγή που έχει γίνει στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά με τον κώδικα συμπεριφορά πρέπει να αναθεωρηθεί, πιστεύετε. Ισχύει από το 2009. Έχουν επέλθει πολλές αλλαγές, η τεχνολογία έχει αλλάξει. Υπάρχουν πιο πολλές επιλογές. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε κανόνες σε μια κατάσταση διαρκώ μεταβαλλόμενη που θα αλλάξει πάλι στο μέλλον. Τι να κάνουμε λοιπόν με μια αγορά που μπορούμε απλώ να προβλέψουμε που ίσω να πάει, προ τα που ίσω να πάει. Να παρέμβουμε εμεί για να τη ρυθμίσουμε. Και φαντάζομαι, κύριε Παγκό, και εσεί ω ε, νέα εταιρεία, νέο νεοφυή, κάτι θα έχετε να πείτε γι' αυτό. Υπάρχει περιθώριο για τι μικρέ νεοφυεί εταιρείε να αναλάβουν κάποιο ρόλο. Είπατε ότι έχετε πολύ μεγάλη δυσκολία να πάρετε χρηματοδότηση και να βρείτε επενδυτέ για να πάρετε χρήμα σε αυτό το τομέα. Ε, να απαντήσουν αμέσως οι προσκεκλημένοι. Εσείς πρώτος. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, ναι, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσουν οι νοαθηφέντες να δραστηριοποιηθούν και να μην ισχύουν οι επιθυντικέ ρήτρε που προστατεύουν του ήρα. Ε, έχουμε εκατοντάδε εταιρείε, ε, δεκάδε εκατοντάδε ταξιδιωτικά πρακτορία. Θα μπορούσαμε να έχουμε και πολλού νέου ε, στην αγορά. Δεν υπάρχει. Ε, δεν θα υπάρχει πρόβλημα όπως τώρα με τη συνάθρηση και θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για τους καταναλωτές ε, σαφέστερη εξήγηση των υπηρεσιών που ε, παρέχονται στους καταναλωτές, όχι μέσω των CRS, και η επιλογή του καταναλωτή θα είναι πιο μορφωμένη, διότι ε, θα έχει καλύτερη εικόνα για το τι του πωλείται. Θέλουμε άλλωστε να μην υπάρχει διάκριση αυτή τη στιγμή μεταξύ των CRS, ε, γιατί ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή σίγουρα πρέπει να υποστεί διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστούμε κύριε Παγκό. Θέλετε κι εσείς να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι μας αφορά, αυτό που έχω να πω είναι ότι κάνουμε, μπορεί να το κάνουν όλοι. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε παίρνουν το API, τις διαπαθές για το σύστημά τους, στην οποία μπορεί να συνδεθεί ο καθένας. Ο GDS, η CRS, Βέβαια για τους GDS είναι κάποιο περίπλοκο το πράγμα γιατί η φιλοσοφία του είναι διαφορετική, η συλλογιστική του είναι διαφορετική σε σχέση με τη διανομή των EPI, αλλά μπορεί να το κάνει κανεί. Το πρόβλημα είναι το χρήμα. Κανεί δεν θα μα δώσει χρήμα. Και η δουλειά που κάνουμε είναι καλή. Αν ρωτήσετε τι αεροπορικέ εταιρείε για την πλατφόρμα μα, έχουν πολύ καλή άποψη. Αν ρωτήσετε του μεταπράτε, ε, την λατρεύουν την πλατφόρμα μα. Την βρίσκουν φανταστική. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει σαφώς πρόβλημα της αγοράς και του κατά πόσον υπάρχει περιθώριο για άλλους. Αλλά το βασικό μας πρόβλημα για μας είναι το ρευστό. Κυρία Ντεμπούστ, και εσείς για την ε, διανομή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Έχετε ρολόι. Πολύ καλά. Θα χρησιμοποιήσω την ε, σύγκριση αυτή και θα αναφερθώ στον πρώην Γενικό Διευθυντή τη American Airlines, τον κύριο Μπράντον πριν από 20 χρόνια. Σε μία διάσκεψη έδειξε απλώς το ρολόι του και είπε «Το πρόβλημα που έχω με την εταιρεία μου είναι πολύ απλό. Εάν θελήσω να βρω τη φθηνότερη τιμή για αυτό το ρολόι στη Νέα Υόρκη, θα πρέπει να πάω σε 2-3 χιλιάδε μαγαζιά. στι αεροπορικέ μεταφορέ, ένα Πελάτη πρέπει να πάει σε ένα πρακτορείο και με μία ενιαία θηρίδα στην ουσία μπορεί μέσω του ταξιδιωτικού πρακτορείου και χάρη στην τεχνολογία GDS μπορεί να δει όλους τους ναύλους που διατίθενται στην αγορά. Αυτό ε, με, ε, πριν υπάρχει να λειτουργεί το διαδίκτυο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ιδίω στα αριστερά μου παρέχουν ε, νέες τεχνολογικές πλατφόρμες και περισσότερη διαφάνεια στον όλο χώρο αυτό, αυτής της αγοράς. Οι αεροπορικές εταιρείε τι λένε. Θα θέλανε λιγότερη διαφάνεια προφανώς και να μην μπορεί να γίνει τόσο εύκολα η σύγκριση. Αυτό ε, έχει να μας διδάξει το unbundling, ο τεμαχισμός των ε, στον άβλο και αυτό είναι και το θέμα του GDS που μας είπε ο κύριος Άουρς ότι είναι θέμα συμφόρησης. Ε, οι ε, εταιρείε αυτές μπορούν να επιβάλλουν τις δικές τους τιμές στην ουσία ε, στις αεροπορικές εταιρείε. Έτσι μας είπε ο κ. Άουρ. Τότε διερωτώ γιατί ο όμιλος Λουφτχάνσα έχει επιφέρει αυτό το πλέον τέλος 16 ευρώ ε, παροχής υπηρεσιών στα εισιτήρια. Θα επηρέαζε αυτό τις πωλήσει της Λουφτχάνσα. Δεν τις επηρέασε. Στις αγορές όπου ήταν δεσπόζουσα η Lufthansa και μιλάω για τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπως προσεκτικοί στο πώ θέτουμε το πρόβλημα. Ναι, εγώ λέω αν είχαμε περισσότερου CRS, αν ήταν περισσότεροι CRS, θα βοηθούσε αυτού του καταναλωτέ για να υπάρχει διαφάνεια. Θα ήταν καλύτερε τιμέ για του καταναλωτέ. Ή υπάρχει εκεί ένα πεδίο, ένας χώρος όπου η διαφάνεια και η έλλειψή της είναι κάτι το επιδιωκόμενο. Εάν εκεί υπήρχε μεγαλύτερος ανταγωνισμός δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Όπως σας είπα, οι νέοι πάροχοι, παρέχοντες, αυτοί παρέχουν νέα τεχνολογικά μέσα, σε ένα βαθμό βοηθούν στην διαφάνεια, αλλά ταυτόχρονα ο εξεβονίμων μου γείτον είπε ότι η δυσκολία είναι από τις χρηματαγορές να πάρει χρήμα. Γιατί? Γιατί τα περιθώρια στις εταιρείες μας αυτή τη στιγμή είναι μακροσκοπικά. Γι' αυτό είναι πολύ μικρά. Γι' αυτό δεν μπορεί ένας επενδυτής να ρισκάρει. Κύριε Βιμ Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνήθω ε, θα πάρω το λόγο στα Ολλανδικά. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν έχουμε πραγματικά ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να ομολογήσουμε και είναι περίπλοκο αυτό το θέμα. Από την παρέμβαση που έκανε ο κύριος Άουερς αντιλαμβάνομαι ότι ε, η δημιουργία αυτών των ε, συστημάτων ε, ουσιαστικά έχει προκύψει από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τώρα. αυτό που κάνετε τώρα ε, είναι η δημιουργία ενός NDC. Καλώς, αλλά γιατί δεν, καταργείτε δηλαδή το σημερινό σύστημα για να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο. Και μετά, ε, ο, αναφέρθηκε ο κύριος στο, στο ζήτημα ε, το, ή μάλλον το, το ζήτημα της ε, χαμηλότερης ε, τιμής αλλά ε, δεν, οι άλλοι ομιλητές δεν αναφέρθηκαν σε αυτό. Εμείς δηλαδή είμαστε κατανοητές που θα κληθούμε στην περίπτωση ενός τέτοιου εντυσσί να πληρώσουμε το κόστος δηλαδή που θα πληρώνουμε σε εσά μετά στην άλλη πλευρά και μετά στην ίδια την αεροπορική εταιρεία για παράδειγμα στη Λουφτκάντσα. Και μετά, στον κύριο Παγκό θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Δεν είσαστε θηγατρική επιχείρηση Αμαντέουσης, δεν είναι. Δεν είστε έτσι θηγατρική της Αμαντέους. Ε, και κύριε ε, Νόλαν, εσείς που εκπροσωπείτε τη Sky Scanner, είστε θηγατρική της Αμαντέους, ούτε κι εσείς. Καλώς. Άρα, Πρόεδρε, εδώ στο Κοινοβούλιο πάντοτε κάνουμε λόγο για τον ανοιχτό ανταγωνισμό και, τις, ε, το δίκαιο ανταγωνισμό. Αλλά όταν κανείς τελικά έχει την, την, τον έλεγχο του 65% της αγοράς, τότε πραγματικά μιλάμε για δεσπόζουσα θέση. Δηλαδή το αμαντέως πραγματικά έχει γιγαντωθεί. Και τι κάνει στο διάμεσο, σύστημα, ε, διάστημα, συγγνώμη, Επιτροπή. Ε, εντάξει, δίνει χρόνο στον εαυτό τη, εξετάζει όλα τα ζητήματα διεξοδικά. Έρχονται τώρα και οι εκλογέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά όλα αυτά μα κοστίζουν χρόνο. Τι να κάνουμε λοιπόν, να επιτρέψουμε για παράδειγμα στον κύριο Παγκό να ε, αποδομήσει την ε, αγορά όπως λειτουργεί αυτή την περίοδο. Ε, ταυτόχρονα η ΆΤΑ είναι πολύ απασχολημένη, οπότε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα. Ξεκινάμε τις απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Διάφορα συγκεκριμένα στοιχεία μας ζητήσατε. Το NDC δεν είναι σύστημα, είναι ουσιαστικά κάτι που προσπαθεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Κάποια πρότυπα ουσιαστικά είναι το NDC με σκοπό να υπάρξει ανταγωνισμός. Η ΑΙΑΤΑ θέλει πραγματικά να αυξηθεί ο αριθμός των CRS δεν μπορούμε να παραμείνουμε με τρία. Δεν μιλήσα για χρήματα. Είπα ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το σύστημα CRS σήμερα. Και για να υπάρξει ελευθερία στη διανομή, για να μην υπάρξουν αυτές οι καταχρηστικές ρίστες, δεν μπορεί εδώ να αυξάνεται το κόστος αναπτύσσει αναεπιβάτη κατά 10 ευρώ. Αυτό είναι υπερβολικό. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη ελευθερία στα δίκτυα διανομής. Τρίτον, Άκουσα ότι είναι πολύ χαμηλή η διανομή. Ναι, εδώ υπάρχει σύγχυση. Είναι πολύ χαμηλές για τους ε, φορείς παροχής υπηρεσιών ή για τις αεροπορικές εταιρείες. Πιστεύω ότι βεβαίως και θα πρέπει εδώ να είναι πολύ διαφανής ε, τα περιθώρια κέρδους στα συστήματα διανομής. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπατε στο τέλος είναι κάτι το οποίο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Πενγκό. Θα ήθελα να πω κάτι που μου φαίνεται καθοριστικό. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στην ε, Lufthansa, στην ε, Air France και σε άλλες αεροπορικές με τον ίδιο τρόπο που συνδέεται με μια πλατφόρμα. Εμείς το κάναμε πολύ απλά. Αν κοιτάξει κανείς, ε, ο καθένας ε, και το Αμαντέος και άλλοι μπορεί να το κάνουν. Δεν είναι μόνο θέμα εμπορικό, είναι και τεχνικό, κυρίως τεχνικό. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Ο τρόπος αυτός, ε, αν θέλετε, μπορεί να αποφευχθεί εάν το σύστημά σας είναι αρκετά σύγχρονο και μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στην αεροπορική εταιρεία. Ναι, Βεβαίω και γίνεται. Έχουμε εταίρους που το κάνουν. Άμεση σύνδεση δηλαδή με τις αεροπορικές εταιρείε. Και ο καταναλωτής αν θέλετε πληρώνει ή πολλές φορές δεν πληρώνει καν κάτι στην πλατφόρμα, στην Skyscanner. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια νέα δομή, έχουμε αυξήσει την εμπιστοσύνη και αυτό είναι η επιτυχία του δικού μας σχήματος. Κύριε Βαντεκάμπ, ε, με το ερώτημα που θέσατε, ουσιαστικά συνοψίσατε τέλεια ε, την ε, εξελίξει κατά τα τελευταία τρία χρόνια στον κλάδο μας. Οπότε σας συγχαίρω. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο ταξιδιωτικό σας ε, ε, πράκτορα στο σπίτι σας ή αν είστε κάτοχος της αεροπορικής εταιρείας. Πραγματικά περιγράψατε πολύ εύστοχα το τι συμβαίνει κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή το GTS καταρχήν ελέγχεται από τις αεροπορικές εταιρείες και εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, υπήρχαν τέσσερα GTS. Γιατί ε, και βέβαια αυτό σήμαινε ότι τα GDS ε, ήταν ε, μεροληπτικά. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι αυτό που κάνουν οι αεροπορικές εταιρείε με τα GDS αποφασίστηκε να αλλάξει το σύστημα. Έτσι λοιπόν το 1989 προέκυψε με αυτό το σκεπτικό ο νέος κανονισμός σε ό,τι αφορά τους κανόνες σε σχέση με την εμφάνιση των διαθέσιμων πτήσεων και ούτω καθεξής. Μετά εδώ ε, κανονισμοί ακολουθούν και τις διάφορες τεχνολογικές ε, ε, εξελίξεις αλλά τη δεύτερη, δεύτερη αναθεώρηση ουσιαστικά αυτό που αποτέλεσαν οι αεροπορικές εταιρείε ήταν να αποεπενδύσουν, δηλαδή να μην επενδύουν πλέον στα GTS και έτσι με αυτόν τον τρόπο βέβαια ήρθαν άλλοι επενδυτές και έχασαν κατά κάποιο τρόπο και τον έλεγχο των GTS και το cash count από αυτές τις δραστηριότητε των GTS. Τώρα τι κάνουν 10 χρόνια μετά θέλουν να επανεφεύρουν ε, το GTS. Πράγμα το οποίο βέβαια θα αποβεί προ ε, ει βάρο και των ε, distributors, δηλαδή εκείνων που προβαίνουν στη διανομή, αλλά και ει βάρο των καταναλωτών. Γιατί όπως είπατε σωστά, ποιο θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό, εγώ και εσεί ω ταξιδιώτε, ω επιβάτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αυτή η πλατφόρμα άμεση σύνδεση, την οποία θέλουν να μα προτείνουν τώρα αεροπορικέ εταιρείε, σε σχέση λοιπόν με αυτή την πλατφόρμα θα μπορούσα, ε, κυρία Πρόεδρε, να σας παρουσιάσω για παράδειγμα μια τέτοια άμεση πλατφόρμα από την πλευρά της ε, Lufthansa και μια, ε, οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα GTS. Και θα δείτε εκεί πολύ εύκολα ποια είναι η διαφορά σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, σε ό,τι αφορά τις ε, προτινόμενες πτήσεις και τις προτινόμενες τιμές. Οπότε ξέρετε τι θα πείτε τότε Πρόεδρε. Για περιμένετε λίγο, προτείνουμε μια τεχνολογία η οποία κινείται πέραν των ορίων της παλιάς τεχνολογίας είναι αυτό που θέλουμε ή θέλουμε να επιμείνουμε στην παλιά τεχνολογία η οποία προσαρμόζεται και η οποία ουσιαστικά υιοθετεί τα πρότυπα ένδυση. Ε, εντάξει, δεν θέλω να μακρηγορήσω ε, κυρία Πρόεδρε, γιατί πραγματικά αρχίζω και ταράζομαι λίγο όταν έχουμε να κάνουμε με αυτήν την, την διανομή εδώ αεροπορικών Ε, Πάντω ε, πραγματικά σα κάνω αυτή την ε, πρόταση κυρία Πρόεδρε, αν θέλει η Επιτροπή σα μία φορά να τη κάνω μία παρουσίαση, ένα live demo, μια επίδειξη δηλαδή live του τι ακριβώ συμβαίνει σε σχέση με, τα διαφορετικά, ε, με τους διαφορετικούς διάβλους του Μαρτίνου και θα δείτε ποιες είναι οι διαφορές. Θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε τέτοια παρουσίαση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόταση. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια σύγκρουση, αλλά εμένα μου το έχουν εξηγήσει. Νομίζω ότι έχουμε ο καθένας από εμά τις δυνατότητες να κατανοήσουμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Στην Αγιάτα εκπροσωπείται όλες τις αεροπορικές και τις μικρές και τις μεγάλες. Έτσι δεν είναι. Όταν όμως κάποιος ουσιαστικά είναι αεροπορική εταιρεία ταξινομείται βάσει του μεγέθους του. Η διανομή λοιπόν εξαρτάται και από το μέγεθος μιας από αεροπορικής εταιρείας. Ερωτώ λοιπόν, οι μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν δικές τους πλατφόρμες. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο για μια μικρή αεροπορική εταιρεία η οποία χρειάζεται είτε τα πρακτορία είτε τις ανεξάρτητες πλατφόρμες πώλησης. Λέτε ότι κάποιες μεγάλες αεροπορικές έχουν ε, ουσιαστικά αυξήσει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων που αγοράζονται μέσω άλλων, ε, αν θέλετε, φορέων, πλατφόρμες κτλ. Τι έχουν κάνει οι μικρές αεροπορικές εταιρείε, Θα σας απαντήσω στα γαλλικά. Το NDC ουσιαστικά είναι ένα σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι αεροπορικές εταιρείε, Ίσες με ίσο τρόπο συγγνώμη για μεγάλες και μικρές. Η ΑΙΑΤΑ δεν είναι ουσιαστικά μια λέσχη για τις ε, μεγάλες μόνο αεροπορικές εταιρείες. Σήμερα έχουν πιστοποιηθεί 60 αεροπορικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες, και μέσω του συστήματός μας ε, ανταλλάσσονται μηνύματα. Ακόμα και μικρές αεροπορικές εταιρείες κατανοούν ότι το σύστημα NDC ουσιαστικά εξυγχρονίζει την ηλεκτρονική της διανομή. Το σύστημα NDC δεν έχει σαν σκοπό να εξαλειφθούν οι ενδιάμεσοι. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν, ε, αν θέλετε, το NDC και τα CRS. Αυτό που είπα είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές ε, συνθήκες για τις αεροπορικές εταιρείες. Το καθοριστικό είναι να υπάρχουν, ε, αν θέλετε, διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης και χειρισμού για τις αεροπορικές εταιρείες. Οι αεροπορικές εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ταξιδιοκτικά πρακτορία. Και εννοείται ότι αυτό θα συνεχιστεί και το, τα γραφεία όπως η Κάλσον και άλλοι σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετούν τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι ένας νέος τρόπος, αν θέλετε, διανομής μέσω του NTC. Και η American Express και η Κάλσον και άλλοι ουσιαστικά χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό γιατί, γιατί τα CRS είτε είναι πολύ αργά, είτε δεν είναι ακόμα ενημερωμένα. Και τα πιο πολλά πρακτορία μας λένε με μεγάλη αγανάκτηση γιατί δεν έχουν ακόμα εξυγχρονιστεί τα συστήματα CRS. Τι έχετε να πείτε σε σχέση με αυτό που μας είπε ο κύριος Άους, κύριε Πενκό. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για την έλλειψη ενδιαμέσων, ουσιαστικά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τη δημιουργία νέων δικτύων. Η δική μας, αν θέλετε, ύπαρξη δικαιολογείται από την δυνατότητα πρόσβασης άλλων, αν θέλετε, φορέων. Η ενσωμάτωση στο GDS είναι πολύ περίπλοκη, στοιχίζει. Υπάρχουν όμως πολλοί οι οποίοι θέλουν να πωλήσουν πτήσεις και σήμερα υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει σύστημα να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να εξαλειφθούν οι ενδιάμεσοι, αν θέλετε. Το NDC δεν είναι το πιο σημαντικό. Το API είναι το σημαντικό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει η διανομή. Η Vueling, η EasyJet και όλες οι, αν θέλετε, εταιρείες προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδεθεί κανείς με αυτούς. Αυτό κάνουν και οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες ουσιαστικά χρησιμοποιούν όλα αυτά τα πρότυπα για να σχεδιάσουν EPIs και μπορεί κάποιος να συνδεθεί κατευθείαν σε μια αεροπορική εταιρεία να συνδυαστεί αυτό με την σύγκριση, αν θέλετε, των πληροφοριών σε μια πλατφόρμα και με την μεταέρευνα να συγκρίνει κανείς σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα. Είναι διαφορετική τρόπη ουσιαστικά σύνδεσης. Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σωστή η ανάλυση σας. Υπάρχουν 240 μέλη της ΑΙΑΤΑ. Περίπου 20 διαθέτουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Οι πιο πολλές περιφερειακές αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη, πολύ σημαντικές για τη σύνδεση κάποιων απομακρυσμένων περιοχών. Έχουμε πάρα πολλές διαδρομές και συνδέσεις από το ένα μέρος στο άλλο και δεν χρειάζεται σαν τις Ηνωμένες να περνάμε πάντα από κάποιες κεντρικές διαδρομές. Είμαστε ένας τομέας ουσιαστικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι πιο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα τέτοιο δίκτυο. Γι' αυτό και ακριβώς επειδή υπάρχουν τα δίκτυα, επειδή υπάρχει το σύστημα front office, back office, λογιστήριο, όλα αυτά συνδέονται. Η δημιουργία νέων προτύπων ουσιαστικά σημαίνει υπερβολικά βαριές επενδύσεις που οι περισσότερες μικρομεσαίες δεν μπορούν να το κάνουν. Θέλετε να πείτε κάτι? Yes, I mean, I think, I think... Ναι. Είναι δίκαιες αυτές οι παρατηρήσεις, σωστές. Υπάρχει σοβαρό κόστος για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουμε. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν ξέρω ποιε είναι οι λύσει που θα βρεθούν στο μέλλον. Τώρα βλέπουμε τι υπάρχει και τι μπορεί να είναι καλό για τους καταναλωτές. Μπορεί βεβαίω να βρεθούν εντωμεταξύ και άλλα καλύτερα και να τακτοποιηθεί από μόνη τη η αγορά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριοι. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Allez, nous continuons. Et je vais Να συνεχίσουμε τώρα. Και θα προσκαλέσω το, τους ε, συμμετέχοντες στο δεύτερο πάνελ. Σας παρακαλώ, ελάτε και λάβετε θέσεις. Alors, je vous les présente. Να σας τους συστήσω. Κύριε Κρουίτ, είστε εδώ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία των Ευρωπαίων Επιβατών. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Κύριε Κλένερ, Γενική Γραμματέα, Ευρωπαϊκή Τεχνολογία και Υπηρεσίες, Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, Ένωση Ευρωπαϊκή Τεχνολογίες και Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών. Και κύριε Ντισάρ, γνωριζόμαστε. Είστε ε, αναπληρωτής διευθυντής της ε, Move. Δεύτερο πάνελ, λοιπόν, Ensuring Neutrality and Transparency λέγεται. Διαφάνεια και ουδετερότητα. Το έχουμε ε, δει κάπως. Υπάρχει κάποιο είδους... Ε, ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών και των ανεξάρτητων πολιτών. Τώρα οι εταιρείε ουσιαστικά μεταπολούν το ίδιο τους το εισιτήριο. Με το πρώτο πάνελ το είδαμε. Είδαμε ότι έρχονται νέες εταιρείε στην αγορά, οι διαδικτυακές πωλήσει εισιτηρίων ή τα CRS, τα Computer Elevation Systems. Τίποτε το απίστευτο και το αδιανόητο, αλλά λίγο να δούμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι δίκαιοι κανόνες για να υπάρχει θεμετός ανταγωνισμός μεταξύ όλων αυτών των ανταγωνιστών. Και εν τέλει να ωφελείται ο καταναλωτής ε, σε κάθε περίπτωση. Ε. Αυτό ε, μας ενδιαφέρει, να θεσπίσουμε νομοθεσία προς όφελος των πολιτών μας για τα εργαλεία αυτά πώληση και κράτηση θέσεων στι ε, αεροπορικέ εταιρείε. Στου τελευταίου μήνε όμω βλέπουμε ένα επιπλέον τέλο από πολλέ αεροπορικέ εταιρείε για τα εισιτήριά του. Γιατί ε, εφόσον εφόσον ανεξάρτητοι τα πράτες ε, τα πολλούν, δεν υπάρχει τέτοιο τέλο, ενώ από την εταιρεία την ίδια απευθεία ναι. Προσφυγή κατά τη Lufthansa έχει ήδη υπάρξει, α πούμε, και κατά άλλων εταιρεών θα έπρεπε να είναι φτηνότερα από τα CRS και αυτό εξαναγκάζει τα ταξιδιωτικά πρακτορία και τους ε, χρήστες να πάνε Από τη στιγμή λοιπόν που οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναπτύξει ένα τμήμα πωλήσεων, θα έπρεπε να είναι και αυτές ένα CRS, όπως όλα τα άλλα. Αυτό θα ήταν το λογικό. Εδώ κάπως ε, προβάλλονται φραγμοί στον ε, θεμητό ανταγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι στο δεύτερο πάνελ, διότι θα θέσουμε τα πραγματικά ερωτήματα που μας ταλανίζουν εδώ. Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερεί εδώ και τρία χρόνια να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Υπάρχει προσφυγή βάσει του κώδικα συμπεριφορά. Γιατί δεν έχει επιληθεί το θέμα, ενώ υποθέσεις είναι τόσες πολλές. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει απορρίψει έστω την προσφυγή αυτή, γιατί οι καταναλωτές μας ρωτούν τι πιστεύουμε. Εξηγούμε ότι ο κώδικας συμπεριφοράς είναι παροχημένος και πρέπει να αναθεωρηθεί πότε θα γίνει αυτή η αναθεώρηση. Αφόσον είναι απριχιωμένο, ε, θα ε, ισχύει δεν θα ισχύει, γιατί δεν έχει αναθεωρηθεί, αναθεωρηθεί αφού είναι τόσο ε, ξεπερασμένο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση ξεκινώντα από το, την καρδιά του θέματο. Διότι από αυτά τα δύο πάνελ θέλουμε να φύγουμε με πραγματικέ συγκεκριμένε προτάσει. Και σα ε, βάζω το. Ε, σα θέτω το πραγματικό πρόβλημα εδώ. Ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τους καταναλωτές. Και πάλι, βάσει των τηρητών του χρόνου, 7 λεπτά έχετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για αυτήν την εισαγωγή. Εδώ παίρνω το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ε, Επιβατών. Δεν βλέπω να εμφανίζεται στην οθόνη ακόμα η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης μου. Ε, εν πάση περιπτώσει, είμαστε μια ε, ε, Ομοσπονδία Διαφορετικών Οργανώσεων με 38 μέλη από 21 κράτη-μέλη. Έχουμε δημιουργηθεί από το 2002 και ουσιαστικά εκπροσωπούμε εδώ την ε, οπτική γωνία των επιβατών ε, στη διάλογο με, τις, ε, με τους διάφορους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό βέβαια στο πλαίσιο και των σιδηροδρόμων και των και της ναυσιπλοείας και των ε, αερομεταφορών. Εδώ βλέπετε τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εγώ ε, ονομάζομαι Άριον Κράουτε και είμαι ε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της Ομοσπονδίας. Ήμουνα ο πρόεδρος της Χόβεν που ήταν η Ομοσπονδία των επιβατών των κάτω χωρών και αυτή ήταν και η δική μου, το δικό μου επάγγελμα. Ε, πρωτού δηλαδή αναλάβω ως μέλος εδώ του, της διοίκησης του EPF και να περάσω τώρα στην παρουσίαση. Τι ακριβώς χρειάζεται ένας επιβάτης. Είναι πολύ απλό. Χρειάζεται αξιόπιστες πληροφορίες σε σχέση με τρία πράγματα. Τα, δρομολο... τα ωράρια δηλαδή των δρομολογίων, ε, το κόστος που είναι διαφορετικό από την τιμή και επίση χρειάζεται αξιόπιστε πληροφορίε ω προ το πώ μπορεί να προβεί στην κράτηση του εισιτηρίου, το booking προτού δηλαδή ταξιδέψει ένας επιβάτης θα προσπαθήσει να ε, βρει αυτές τις πληροφορίες, δρομολόγια, κόστος και τρόπος κράτησης. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα. Υπάρχουν ε, τμηματικές μόνο ε, πληροφορίε σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια. Για παράδειγμα, εγώ θα πρέπει να ταξιδέψω στον επόμενο μήνα από το Άμστερνταμ στο Όσλο. Κανονικά ε, πρόκειται για ένα πολύ απλό δρομολόγιο. Αν θέλω να μάθω τι ώρε, ε, θα πρέπει να πάω στην KLM και θα ενημερωθώ σε ό,τι αφορά τι ημερήσιε πτήσει. Μετά θα πάω στο site τη SAS, θα με ενημερώσουν σε ό,τι αφορά τι ημερήσιε πτήσει του και μετά θα πάω σε μία από αυτές τις ε, ιστοσελίδε, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες από τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αλλά όχι από όλες γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις δεν έχουν τις πληροφορίες από ε, από όλου του αερομεταφορεί, για παράδειγμα, συχνά σε τέτοιου είδου πλατφόρμε δεν περιλαμβάνεται η Ryanair, ενώ σε άλλε δεν περιλαμβάνεται η EasyJet. Οπότε θα πρέπει ε, να δούμε εκεί, να δει κανεί ποιε είναι οι εναλλακτικέ. Μετά τα πράγματα γίνονται ακόμα περίπλοκα σε ό,τι αφορά το κόστο. Και επαναλαμβάνω, το κόστο είναι διαφορετικό από την τιμή. Ε, δηλαδή, ξέρουμε όλε αυτέ τι διαφημίσει που λένε μπορεί κανεί να πάει από το Άμστερνταμ στο Όσλο ξεκινώντα από τάδε τιμή, αλλά και βέβαια η τιμή είναι αστεία, είναι εξαιρετικά χαμηλή, αλλά δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά το κόστο ε, και υπάρχουν τα συμπληρωματικά, οι συμπληρωματικέ χρεώσει και τα ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Δηλαδή υπάρχουν συμπληρωματικέ ε, επιβαρύνσει, τι οποίε δεν γνωρίζω. Υπάρχουν συμπληρωματικέ δαπάνε σε ό,τι αφορά ε, τι αποσκευέ και είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα εδώ γιατί πληρώνει κανεί επιβάρυνση σε ό,τι αφορά 10 κιλά ή κιλά, 20 κιλά, 23 κιλά ή 30 κιλά. Οπότε πρέπει κανεί να κάνει μια ολόκληρη έρευνα για να μάθει τι καλύτερα να καταβάλει. Και ορισμένες περιπτώσεις ε, δείχνουν ότι ε, το ειστήριο είναι πιο ακριβό ή το κόστος σε ό,τι αφορά την αποσκευή παρά για τον ίδιο τον επιβάτη. Και μετά έχουμε τα, ε, επιπρόσθετα, το επιπρόσθετο κόστος σε ό,τι αφορά την ε, την κράτηση δηλαδή. Ε, χρησιμοποιούν πολύ ε, Ολλανδοί το IDO και αν δεν μπορεί όμως κάποια στιγμή να έχει πρόσβαση στο IDO θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ε, την πιστοτική του κάρτα και αν χρησιμοποιήσει την πιστοτική κάρτα θα πρέπει να καταβάλει ένα τέλος για τη χρήση της πιστοτικής κάρτας για την κράτηση. Και μετά υπάρχουν και ε, το, οι κρυφές δαπάνε, το κρυφό κόστος γιατί συχνά πρέπει να ταξιδέψουν από το ένα σημείο στο άλλο, όχι από ένα αεροδρόμιο στο άλλο. Άρα λοιπόν θα πρέπει εγώ καταρχήν για παράδειγμα αν θέλω να πάω από το Άμστερνταμ στο Όσλο θα πρέπει να πάρω από το Άμστερνταμ έως το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ένα ε, τρένο ή ένα αυτοκίνητο και μετά. Όταν θα φτάσω στο Όσλο δεν πρέπει να βέβαια μείνω στο αεροδρόμιο, θα πρέπει να φτάω ε, να πάω σε ένα ε, προάστιο του Όσλο. Πώ θα συνεχίσω το ταξίδι μου. Μπορώ να συνεχίσω με ένα ταξί, το οποίο μάλλον θα είναι πάρα πολύ ακριβό, ή μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα λεωφορείο. Αλλά πού βρίσκεται η στάση του λεωφορείου και πώ θα πληρώσω για το ειστήριο του λεωφορείου στο, Όσλο. Ε, στο Όσλο. Δεν έχω ιδέα. Μετά, μπορώ να πάρω ένα τρένο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά τρένα. Υπάρχει το φλέκτοκα το οποίο είναι πολύ καλό, πολύ άνετο, αλλά είναι πολύ ακριβό και μετά έχω ένα τρένο ε, της δημόσιας επιχείρηση σιδηροδρόμων, το οποίο ε, δεν είναι τόσο καλό, αλλά είναι πιο φτηνό ε, και μου δίνει ένα εισιτήριο που ισχύει για το σύνολο του όσο. Αλλά πώς μπορώ να μάθω λοιπόν όλα αυτά τα ε, κρυφά ε, κόστη, τι κρυφέ δαπάνε. Γιατί βέβαια αυτά είναι που επηρεάζουν την τελική τιμή και όχι μόνο η τιμή του ειστήριου αυτού καθεαυτού. Ε, και εδώ λοιπόν έρχομαι σε αυτό που θα θέλαμε να λαμβάνουμε ω επιβάτε. Καταρχήν, πληροφορίε σε σχέση με όλου του αερομεταφορεί και εύκολη πρόσβαση ε, σε αυτέ τι πληροφορίε για να ξέρουμε πού μπορεί κανεί να κάνει μια κράτηση και πού μπορεί να βρει τι ειδικέ πληροφορίε. Θέλουμε επίση διαφάνεια σε ό,τι αφορά το κόστο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρη αδιαφάνεια προ το τι πληρώνουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχουν διαφορέ στο των τιμών στους διαφορετικούς διάβλους διανομής. Δηλαδή αυτή η επιπρόσθετη, το επεισόδιο τέλος από την πλευρά του Λουφχάντσα είναι κάτι το πολύ κακό και φοβούμε ότι αν δεν αναλάβει δράση η Επιτροπή θα αρχίσει να εξαπλώνεται κι αλλού. Και ένα τέταρτο σημείο το οποίο νομίζω πως θα εκτιμήσετε, είναι το ότι θέλουμε να έχουμε την πληροφορία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Βλέπουμε το, ε, πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δραστηριοποιείται πάρα πολύ σε αυτό το τομέα και είμαστε ευγνώμονες, αλλά πόσοι πραγματικά γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Εάν για παράδειγμα κάνω μια κράτηση σε ένα ταξιδιωτικό πράκτορα και υπάρχει σε ένα πρόβλημα. Πού πρέπει να απευθυνθώ, στον ταξιδιωτικό πράκτορα, στον αερομεταφορέα. Δεν το γνωρίζω. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση των επιβατών σε ό,τι αφορά όχι μόνο τα δικαιώματά του, αλλά και την πρόσβαση στα δικαιώματά του, την άσκηση των δικαιωμάτων. Και όπω είπα και προηγουμένω, θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίε σε ό,τι αφορά το ταξίδι πέραν του αεροδρομίου που δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο στο σύνολο των αερομεταφορών και δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ωραία. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον δεύτερο προσκεκλημένο μας. Στον κύριο Κλένερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που υποδέχεστε. Ε, με πιάνει μια νοσταλγία, γιατί θα είναι η, προ... η τελευταία μου δημόσια εδώ μετά από 9 χρόνια στην την θέση. Ε, ήταν χαρά μου να συνεργάζομαι με το Κοινοβούλιο και θα παρακολουθώ τις εργασίες σας στο μέλλον. Αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα βάσει των όσων προβλέπει το πρόγραμμα εργασιών. Εγώ εκπροσωπώ την ΕΤΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Εταιριών ε, ταξιδιωτικών τεχνολογιών. Θα ξέρετε πολλές από αυτές ε, που βλέπετε και στη διαφάνεια. Και σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στον κώδικα συμπεριφοράς των CRS. Γιατί υπάρχει, ποια είναι η αξία του και από τη δική μας την προοπτική ποιο θα έπρεπε να είναι το μέλλον. Εάν μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Όπως είπε και ο κύριος Φάντενκαμπ σωστά, οι αεροπορικές εταιρείες δημιουργήσαν τα CRS αρχικά τη δεκαετία του 70 και του 80. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να απορριθμίσει τον τομέα των αερομεταφορών, είπαν ότι χρειαζόμαστε εγγυήσεις για τον ανταγωνισμό για να μπει κανεί στην αγορά και για του καταναλωτέ. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο κώδικα συμπεριφορά των CRS. Για να αποτρέψει τι αεροπορικέ εταιρείε από το να ε, ε, επεκτείνουν την δεσπόζουσα, την δεσπόζουσα θέση τους. και να μπορεί να υπάρξει και άφηξη, έλευση νέων ανταγωνιστών. Ε, ο κώδικας συμπεριφοράς έφερε ουδετερότητα και διαφάνεια της, ε, στην ενημέρωση, οπότε υπήρξε δυνατότητα να έρθουν και νέοι ανταγωνιστές, να παίξουν περισσότερες πληροφορίες και να χαμηλώσουν τιμές για τους καταναλωτές. Άκουσα σχόλια για το κόστος διανομής αυτή τη στιγμή στη σημερινή συζήτηση. Υπάρχει μια ανεξάρτητη μελέτη από μια εταιρεία που λέγεται Φράλτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκανα την κοπιώδη δουλειά να συγκρίνει το κόστος της άμεσης διανομής των εισιτηρίων και κάτι που δεν μας εξέπληξε μεταξύ των πορισμάτων είναι ότι η έμεση διανομή είναι αποτελεσματικότατος τρόπος πώλησης περιεχομένου. Και έχει χαμηλότερο κόστο σε σύγκριση με την άμεση πώληση. Να σα πω και το άλλο. Όταν μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία που όλοι γνωρίζουμε ε, έφτασε να δικαστεί στην Αυστρία για το ε, διαβόητο επιπλέον τέλος έπρεπε να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν δικαιολογημένο το επιπλέον αυτό κόστος. Μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να υποβάλουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Κάτι που πραγματικά είναι κάτι που μας ε, κλείσει. Ε, επόμενη διαφάνεια. Τα τελευταία 10-15 χρόνια με την ανάδυση του διαδικτύου, τη διάδοσή του και τη χρήση του από όλου του καταναλωτέ σχεδόν, βλέπουμε νέους διάβλους διανομής. Κάποιοι είναι ρυθμισμένοι, κάποιοι όχι. Και κάποιοι είναι προφανώς ε, μεικτοί. Είναι οι διάβλοι που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείε ε, υπογείως. Ε, εδώ λοιπόν οι σχέσεις μεταξύ τους είναι πολύ σημαντικές. Σήμερα ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 50% της διανομής των αερομεταφορών και των υπηρεσιών τους να πηγαίνουν απευθείας ε, και όχι στα ταξιδιωτικά πρακτορία και τους ε, πρακτόρες. Είναι νομίζω περιβολή όμως να μιλάμε για σημεία συμφόρησης. Μιλήσαμε για το επιπλέον κόστος τα ε, επιπλέον αυτά είναι σύμπτωμα ενό ευρύτερου προβλήματος και αυτό έχει να κάνει με την διάκριση του, διεύλου, του διάβλου. Ε, μπορεί να, να έχει να κάνει και με την ε, διάκριση του περιεχομένου που διατίθεται από τον κάθε διάβλο διανομής. Θα μπορούσε κανείς να πει δεν είναι ελευθερία επιχειρηματική μια εταιρεία να αποφασίσει με ποιον θα ε, κάνει business, σε ποιον θα δίνει περιεχόμενο και σε ποιον θα πουλάει τα προϊόντα της. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη, σίγουρα. Αλλά είναι δύο οι όψεις του νομίσματος της αγοράς. Από την άλλη πλευρά ε, κάθεται και ένας καταναλωτής, τον οποίο δεν τον εξυπηρετεί σε τίποτα κατακαιρματισμός. Θέλει να μπορεί σε ένα σημείο να συγκρίνει όλες τις προσφορές που υπάρχουν, διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνει μια μορφωμένη επιλογή. Και η άλλη πλευρά, ο άλλος δρόν στην αγορά, να είναι κάπως πειθαρχημένο πώς να ανθεί ο ανταγωνισμός στις αερομεταφορές εάν δεν υπάρχει καμία πειθαρχία και καμία διαφάνεια. στις μεικτές πλατφόρμες, με τη διάκριση των διάβλων, με τις προκαταλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, αυτό προκαλεί ένα μεγαλύτερο μέρος ε, της αγοράς ε, να είναι στα χέρια κάποιων λίγων αερομεταφορέων. Κάτι που πλήττει τον ανταγωνισμό. Αυτό το είδαμε ήδη να συμβαίνει. Αεροπορικέ εταιρείε που έχουν δεσπόζουσα θέση την ενισχύουν με διαφορετικούς τρόπους. Μεταξύ άλλων και με τη διάκριση των διάβλων θα είναι δυσκολότερο για του καταναλωτέ να συγκρίνουν μέσω αυτών των διάβλων, διότι ο κατακαιρματισμό δεν είναι κάτι το καλό. Και να είμαι ξεκάθαρο, ένα καταναλωτή αποφασίσει να αγοράσει από έναν διάβλο απευθεία από μια αεροπορική εταιρεία, είναι επιλογή του. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν όμω δυσκολεύεται τον καταναλωτή να συγκρίνει, για αυτού που θέλουν να συγκρίνουν, και κατά την άποψή μου και φαντάζομαι ότι Άρια θα συμφωνήσει, έχουν δικαίωμα να συγκρίνουν, αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Εάν μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια, πολύ συγκεκριμένα για τις προσφυγές ε, που έχουν ε, υποβληθεί πριν από τρία χρόνια περίπου κατά της Λουφτκάντζα, για, τον για το διαβόητο επιπλέον κόστος. Ξέρω, Κριστόφ, ότι έχετε πολιτικούς προϊσταμένους, οπότε μην το πάρετε ως κριτική, αλλά πραγματικά είναι ε, κάτι που προκαλεί έκπληξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και τρία χρόνια δεν έχει αποφαλθεί για τις προσφυγές αυτές και δεν τις έχει απορρίψει καν να είμαστε σαφείς. Έχει αποφασίσει να μην εφαρμόσει τους κανόνες. Διότι εντωμεταξύ μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να αλλάξουν οι κανόνες. Εάν αυτό γίνει η νέα πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι η επιβολή της νομοθεσίας γίνεται κάτι το περιττό. Τι καθόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε. Γιατί σχεδιάζουμε νόμους άμα δεν χρησιμοποιούνται και δεν εφαρμόζονται. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεταβάλει τη στάση τη και να πάρει λίγο σοβαρά τους κανόνες που ισχύουν. Ο κανονισμό είναι σε ισχύ. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί μέχρι να αναθεωρηθεί. Και πολύ σύντομα, ε, έχω τρει σύντομε παρατηρήσει παρόλο που έχω ξεπεράσει το χρόνο μου για το μέλλον του κώδικα συμπεριφορά ή όπω ονομαστεί τέλο πάντων. Μπορεί να του δώσουν άλλο τίτλο θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τους νέους διάβλους διανομής που έχουν δημιουργηθεί. Να δει πολύ καλά το σημερινό τομείο διανομής και να σκεφτεί ίσως και το μελλοντικό προσπαθώντα να διασφαλίσει την ουδετερότητα, τη διαφάνεια και την πρόσβαση στι πληροφορίε για του καταναλωτέ. Και, όπω είπα και προηγουμένω, ποιο είναι το νόημα τη νομοθεσία, αν η νομοθεσία δεν επιβάλλεται, δεν εφαρμόζεται. Ο ισχύον κώδικα και οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία στον χώρο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται. Θα πρέπει να επιβάλλεται εν ευθέτω χρόνο για σκοπούς νομικής ασφάλειας και για όλους τους ε, δρόντες στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Κλένερ και τελευταίος μας ε, προσκεκλημένος ο κύριος Δισάρ για 7 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να πάρω το λόγο εδώ στα πλαίσια αυτού τη συζήτηση, ένα θέμα που μας αφορά όλους. Έχω και εγώ λίγο χρόνο, οπότε θα περιοριστώ στο δικό μας, αν θέλετε, όραμα, πώς βλέπουμε την προσέγγιση τη δική μας για τον κώδικα συμπεριφοράς μετά την τελευταία αναθεώρηση και μετά την αξιολόγηση που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 βάση των κανόνων διαφάνειας των τιμών που αφορά το κείμενο αυτό. Τον Οκτώβριο του 2015 δημοσιεύσαμε έναν οδικό χάρτη μετά από μια πρώτη ανάλυση που κάναμε όσον αφορά τα διάφορα θέματα που θέλαμε να αξιολογήσουμε και μετά από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση για ένα χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 κάτι που ουσιαστικά αποτελεί μια συμπληρωματική, αν θέλετε, δραστηριότητα σε σχέση με όλα όσα έχει κάνει η Επιτροπή προηγουμένως, ανταλλαγή απόψεων με τους υπεύθυνου κτλ. Το Μάρτιο του 2017 ξεκίνησαν τα πρώτα συμπεράσματα να παρουσιάζονται και να δημοσιεύονται και η ιδέα να ξεκινήσει ένα καινούριο κείμενο και βεβαίως ε, ουσιαστικά ξεκινήσαμε με, την προηγούμενη, με το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ολοκληρωθεί όμως η αξιολόγηση και θα παρουσιαστεί το νέο κείμενο με το νέο Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Συνεχίζουμε τις ε, αξιολογήσεις ε, παρακολουθώντας τα δεδομένα της αγοράς και οι προτάσεις μας ουσιαστικά λαμβάνουν υπόψη όλη την καινοτομία των δικτύων διανομής, κάτι που μας οδηγεί σε νέο κείμενο. Είναι πολύ νωρίς βεβαίως να σας δώσω τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης, γιατί βρισκόμαστε στην αρχική φάση, αλλά ακούγοντας αυτά που υπόθηκαν εδώ σήμερα το απόγευμα και βάσει των πρώτων επαφών που έχουμε με τους εμπλεκόμενους φορείς του τομέα, θα ήθελα να σας πω ότι πρώτον, στο σύνολο του τομέα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα δίκτυα διανομής τους. Αυτό είναι μια γενική αρχή την οποία θέλουμε να τηρήσουμε. Δεύτερον, μας φαίνεται σαφές ότι όλοι οι φορείς στην αγορά θα πρέπει να υπακούν τους ίδιους κανόνες. Και το Travelport και το SAM και το Amadeus ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Υπάρχουν όμως και άλλοι, αν θέλετε, εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι ακολουθούν άλλους κώδικες συμπεριφοράς και ιδιωτολογίες και αυτό θα πρέπει εδώ να ε, εναρμονιστεί και είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει σαν προτεραιότητα. Σήμερα το απόγευμα είδαμε ότι πραγματικά ο καταναλωτής βρίσκεται στο κέντρο της ε, προσπάθειάς μας και σε μας στην ε, Επιτροπή. Ο καταναλωτής μπορεί σήμερα, και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, να συγκρίνει τις τιμές, την παροχή υπηρεσιών, τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει άρθρο 5 του σημερινού κανονισμού απαιτεί από όλες τις ε, επιχειρήσεις ουδέτερη αναφορά, χωρίς διακρίσεις. Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί, θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όπως είπε ο κύριος Λενέρ, η αξιολόγηση αυτού του κώδικα συμπεριφοράς ουσιαστικά συμβαίνει σε ένα περιβάλλον ε, συγκεντρώσεων ε, και εξαγορών από μέρος των αεροπορικών εταιριών, κάτι το οποίο είναι μια τάση που συνεχίζεται και θα συνεχιστεί στο μέλλον. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να παραμείνει ο ανταγωνισμός αθέμητος γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ε, ο καταναλωτής να μην μπορεί να συγκρίνει τα στοιχεία που τους παρουσιάζονται. Συνεχίζουμε λοιπόν την εξέταση όλων αυτών των ε, προτάσεων και βεβαίως θα συνεχιστεί η υπερξεργασία και η συζήτηση και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντουσάρ. Ξεκινάει η συζήτηση αμέσως. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας. Περίπου τις ίδιες ερωτήσεις με το προηγούμενο πάνελ θα έχω, κυρίως για τον κύριο Τισάρ της Επιτροπής. Ήθελα να μου πείτε προσφυγές από προμηθευτές για το επιπλέον τέλος έχουν υποβληθεί. Το ξέρουμε αυτό κατά τα 6 ευρώ και το επιπλέον τέλος. Και βλέπουμε να διαδίδεται ως ασθένεια και σε άλλες αεροπορικές. Κατάλαβα ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή αναθεώρηση. Γιατί όμως δεν χρησιμοποιείτε τον τωρινό κώδικα συμπεριφοράς για να ασχοληθείτε με την προσφυγή. Μα είπατε ποιο είναι ο δικό σα χάρτης, α πούμε, για τι διαβουλεύσεις το 2019, ότι δεν θα γίνουν όλα αυτά μέσα στη θητεία αυτή. Δεν θα έχει συσταθεί σε σώμα για ένα διάστημα το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα αλλάξει. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, πολύ χρόνο. Μπορεί να φτάσουμε 2019 και αρχές 2020 μέχρι να ξανασυναντηθεί, να ξανασυνέλθει αυτή η Επιτροπή. Αυτό το επιπλέον λοιπόν κόστος και εφόσον διαδοθεί και σε άλλες εταιρείες, ε, ουσιαστικά βαρύνει τον καταναλωτή. Αυτοί το πληρώνουν οι καταναλωτές. Εξηγήστε μου λοιπόν λιγάκι γιατί δεν κάνατε τίποτα βάσει του ισχύοντος κώδικα συμπεριφορά. Και για τον κύριο Κλένερ. Για το επιπλέον τέλος. Πού πηγαίνει αυτό ο καταναλωτής τελικά το επιβαρύνεται. Για λόγους διαφάνειας είναι κάτι που μας ανησυχεί. Διότι θα μπορούσαμε κάπου να συζητήσουμε και κάτι άλλο, Ας πούμε, με τα αεροδρόμια για τι αεροπορικέ εταιρείε τι γίνεται. Ποιο πληρώνει εκεί την πλέον τέλεια. Αλλά τέλος πάντων οι καταναλωτέ είναι αυτοί που ουσιαστικά το πληρώνουν. Ευχαριστούμε κυρία Κλούν. Κυρία Ταπαρδέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, συμμετέχοντες σε αυτό το πάνελ. Οπωσδήποτε θα θυμούνται οι συνάδελφοι μεταξύ αυτών που έχουν εντοπίσει αυτό ακριβώ το πρόβλημα, το επιπλέον τέλο που επιβάλλουν κάποιε αεροπορικέ εταιρείε. Είναι πραγματικά μια πρακτική που υπονομεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και αντίκειται στο, ε, στην αρχή τη διαφάνεια ό,τι αφορά το κόστο ενό ταξιδιού. Επιπλέον, είναι απειλή κατά τη ε, ανταγωνιστικότητα και τη έννοια αγορά των αερομεταφορών. Δημιουργείται ανταγωνισμό ω προ τι τιμέ τελείω τεχνητό και πραγματικά αυτό βλάπτει τους καταναλωτές. Είμαστε σε μια ενιαία αγορά, ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Ο καταναλωτής θα έπρεπε να μπορεί να ενημερώνεται, να συγκρίνει ε, στο διαδίκτυο τις προσφορές και το κόστος. Όμως τη στιγμή που αγοράζει ένας καταναλωτής το εισιτήριό του, ε, πώς ξέρει τι ακριβώ πληρώνει με αυτόν τον ταμαχισμό των αποσκευών, του ναύλου και το καθεξής. Δυστυχώ οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν επαρκώ. Και πραγματικά η κατάσταση αυτή ε, είναι τελείω αντίθετη με τα όσα προβλέπει ο τωρινό κώδικας συμπεριφορά. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αναθεωρηθεί ο κώδικα συμπεριφορά, αλλά με τότε τι θα γίνει. Θα πρέπει να ε, αλλάξει η κατάσταση αυτή στο μέλλον. Ίσως να υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφορά που θα, θα, θα δώσει λύσεις, αλλά δεν είναι αυτό απάντηση για να καταναλωτή σήμερα. Θα πρέπει να λάβουμε κάποια στιγμή κάποια απάντηση. Στι γραπτέ με ρωτήσει δεν έχω λάβει καμία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τι θα κάνει για να διασφαλίσει ότι υπάρχοντε κανόνε γίνονται σεβαστοί. Εδώ πραγματικά υπάρχει έλλειψη ε, απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό εμέσω δεν θα ερμηνευόταν ω υποστήριξη των πρακτικών αυτών. Πρακτικών που όμω ε, υπονομεύουν τη διαφάνεια, υπονομεύουν του καταναλωτέ οι πρακτικές αυτές δεν είναι ένα προηγούμενο αρνητικό για οποιοδήποτε που παρέχει υπηρεσίες και όχι μόνο στις αερομεταφορές. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι επιβάτε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των αερομεταφορών και τι διανομήσει των υπηρεσιών του, χωρί να πρέπει να ε, πληρώνουν ένα επιπλέον κόστο δεν μιλάμε για έναν μικρό αριθμό επιβατών, μιλάμε για εκατομμύρια ταξιδιώτες στην Ευρώπη. Είναι εκατομμύρια οι πελάτες και οι καταναλωτές που χάνουν χρήματα και τους επηρεάζουν όλα αυτά. Πού πάει αυτό το χρήμα, χάνεται. Εμεί, ω Ευρωπαίοι νομοθέτε, έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Εμεί ευχαριστούμε, κυρία Ταπραντέλ. Κύριε Ρικέ, δεν ζητήσατε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της α, βραδύτητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λέω και δεν τους να μου εξηγήσετε γιατί. Επί τρία χρόνια η DG Move εξετάζει τις προσφυγές το CRS 80-2009 Και τελικά ουσιαστικά απορρίψατε ότι η Λουφτχάνσα έχει δράσει παράνομα. Λέτε την ίδια ώρα ότι είναι απαρχαιωμένος ο κώδικας συμπεριφορά κτλ. κτλ, κτλ. Σας παρακαλώ, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Ακούστε με, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί όταν ο καταναλωτής αντιμετωπίζει δυσκολίες, στρέφεται προς εμάς, τους νομοθέτες. Και τι μας λέει, τι κάνατε για να με προστατεύσετε. Όλοι εδώ σε αυτή την επιτροπή ουσιαστικά προστατεύει μία βασική αρχή της ψηφιακής διανομής που είναι η ουδετερότητα. Οι σχέσεις λοιπόν μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και των CRS Computer Reservation System, ουσιαστικά θα πρέπει να διασφαλίσει αυτήν την ουδετερότητα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερο, όσον αφορά τις προσφυγές που έγιναν από μέρους του OTTSA το 2015 κατά του ομίλου Lufthansa. Επαναλαμβάνω, είναι επίγον το θέμα. Γιατί κάνατε τρία χρόνια να εξετάσετε αυτό το θέμα. Είναι κατεπίγουσα υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος θεωρεί ότι έχουν πληγεί τα συμφέροντά του, πρέπει κάτι να κάνουμε. Η τελευταία μου ερώτηση απευθύνεται κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποιο βαθμό και με τι ταχύτητα θεωρείτε ότι μπορεί πραγματικά να αναθεωρηθεί αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς που εσείς οι ίδιοι θεωρείτε ότι είναι απαρχαιωμένος και πεπερασμένος. Και πείτε μου, ξεπερασμένος, συγγνώμη, και πείτε μου, ε, από τη στιγμή που είναι απαρχαιωμένος, γιατί δεν δράτε ταχύτερα. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα δώσω λοιπόν το λόγο σε όλους, εδώ στο πάνελ, και θα απαντήσει πρώτα η Επιτροπή. Είστε ένας από τους υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ άμεση η ερώτηση που μου κάνετε και θα απαντήσω κι εγώ πάρα πολύ άμεσα. Όσον αφορά τις προσφυγές που έχουν ε, υποβληθεί κατά της ε, Lufthansa για το επιπλέον κόστος, πήρε χρόνο η υπόθεση αυτή, ήταν περίπλοκο τα κείμενο, Ήταν περίπλοκη επίσης η εξεχνίαση της υπόθεσης αυτής και φτάσαμε σε κάποια, αν θέλετε, προκαταρκτικά συμπεράσματα, τα οποία έχουμε υποβάλει. Συνεχίζουμε όμως την εξέταση του θέματος αυτού και θα υποβάλουμε τα τελευταία μας συμπεράσματα. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι εν εξελίξη, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω για το σημείο αυτό όπως έλεγε ο Γενικός Διευθυντής, ξεπερνάει, αν θέλετε, τις δυνατότητές μου και τις δυνατότητες που προσφέρει η θέση μου. Και εγώ να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Κλούν. Λέτε, ουσιαστικά ρωτάτε ποιος πληρώνει. Ο καταναλωτής, ο χρήστης. Μία απλή μαθηματική άσκηση είναι αυτή κοιτάξτε ότι μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία αλλά και άλλες ουσιαστικά αεροπορικές εταιρείες, πέρα δηλαδή από τον γνωστό γερμανικό όμιλο, ο οποίος επιβάλλει αυτό το επιπλέον κόστος. Ουσιαστικά, επί τρία χρόνια βλέπουμε, και αυτό είναι δημόσια στοιχεία, από την ετήσια έκθεσή τους. Αν πάρετε τον αριθμό των ε, εισιτηρίων επί 50% επί 2, γιατί ουσιαστικά ένα στα στήρια περνάει μέσω των ανεξάρτητων ε, σημείων πώλησης. Επί 16 βλέπετε το ποσό. Ήταν πάρα πάρα πολύ δημιουργική αυτή η εφεύρεση. Πάνω από ένα δις ή σχεδόν ένα δις είναι το ποσό ουσιαστικά που ουσιαστικά μπήκε στα ταμεία του ομίλου αυτό, της Lufthansa, ένας πολύ δραστήριος όμιλος στην Ευρώπη, χάρη σε αυτό το επιπλέον κόστος των 16 ευρώ. σε ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Yes, I think it's quite right. It is in the Νομίζω πως ε, είναι σωστό αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι το συμπληρωματικό τέλος το καλύτερα να το πληρώσει ο, επιβάτες και αν κάνει κανεί ε, άμεσα μια κράτηση στην KLM ή στη Lufthansa ή σε ένα έμεσο κανάλι, θα διαπιστώσει ακριβώ τη διαφορά που υπάρχει στην τιμή και το συμπληρωματικό τέλο. Αλλά δεν είναι τόσο έξυπνοι όλοι οι καταναλωτέ. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καταναλωτέ, πάλι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ε, δεν γνωρίζουν ακριβώ ε, πώ να ψάξουν και να βρουν την καλύτερη τιμή που υπάρχει στο διαδίκτυο. Και εμεί θα θέλαμε λοιπόν να συνεχίσει ο σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορε. Έχουν παίξει ένα σοβαρό ρόλο ακόμα και την εποχή του διαδικτύου, ειδικότερα για του επιβάτε οι οποίοι ε, δεν έχουν ε, τόσο καλή εξοικείωση με το διαδίκτυο και δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για το γεγονό ότι δεν είναι τόσο καλά εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλε ερωτήσει. Εγώ έχω μια ερώτηση. Εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι προσωπικό, κύριε Ντουισάρ, αλλά συμφωνώ με την κυρία Ταπαρντέλ. Μας λέτε δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση γιατί ξεπερνά το δικό μου το μισθό και την θέση μου. Ε, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εμείς όμως χρειαζόμαστε απάντηση. Ε, αυτή τη στιγμή ε, εκπροσωπούμε πολίτε, ε, κάποια στιγμή πρέπει να μπορούμε να του λογοδοτήσουμε. Και εκείνον ε, του έχουν λίγο βάλει χέρι. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Κύριε Ντισάρ, θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την κυρία Ταπαρντέλ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντουισάρ που ήρθατε και συμμετείχατε σε αυτό το πάνελ. Σας ευχαριστούμε και εσάς κύριε Κρούτ και κύριε Κλένερ. Σας χειροκροτούμε και ευχαριστούμε που μας αφιέρωσετε χρόνο. Είναι ένα θέμα που απλώς αρχίζουμε να εξετάζουμε το ή άλλω. Madame Ε, λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας. Ε, συνεχίζουμε με την έκθεση Ζήλε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζήλε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζήλε που επιτρέψατε να αναβληθεί η εξέταση του θέματό σας. Αρχικά να καλωσορίσω μια νεαρά, μια πολύ μικρούλα, δίπλα στην κυρία Βιέ. Πώ σε λένε, Καμίγ, έλα Καμίγ δίπλα μου στο προεδρείο έλα να προεδρεύσουμε μαζί σε αυτό το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης. Χειροκροτήματα για την Καμίγ. Madame Vieux, elle peut venir à côté de moi? Oui. Έλα, μπορεί να έρθει δίπλα μου. Ωραία. Πόσο είσαι, Καμίλη. Δέκα και μισό. Είσαι έτοιμη? Λέει όχι. Τώρα είναι έτοιμη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε <laughs> τη συνεδρίαση. Μπράβο, Καμιγέλα, πιο μπροστά. Ανοίγει το μικρόφωνο και λε καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Oh! Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Πολύ γλυκούλα. Λοιπόν, ξεκινούμε. Δεν ξέρω αν θα καταλάβει όλη σα την έκθεση, κύριε Ζήλε αλλά να ξεκινήσουμε με την ε, πρόσβαση στις ε, διεθνείς αγορές για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Συμπρόεδρε. Τα λεωφορεία και τα πούλμαν ήταν ένας από τους σημαντικότερους τρόπους μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ε, ε, αστικές περιοχές των κρατών μελών και αποτελούν το μόνο τρόπο μετακίνησης σε ορισμένε από αυτές τις περιοχές αλλά και τις υπαίθριε περιοχέ, και γι' αυτό είναι σημαντικό οι επιβάτες μας να λαμβάνουν ποιοτικέ υπηρεσίε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης. Όταν ένας μεταφορέας που θέλει να εισέλθει μέσα ε, στην, αγορά ενός κράτους ε, μέλους να μπορεί να παρέχει τι υπηρεσίες του περιφερειακά χωρί να υπάρχει κάποιο εμπόδιο, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ισχύει σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, δηλαδή, ε, κάποιοι ανέφεραν συνάδελφοι ότι πρόκειται για ένα καλό καμποτάζ, δηλαδή σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχει κακό καμποτάζ, ενώ εδώ υπάρχει ένα καλό καμποτάζ και νομίζω πω αυτό είναι ο βασικό στόχο αυτή τη έκθεση. Ε, οι δικοί μου συνεργάτε λοιπόν ε, εργάζονται από αυτού του φακέλου. Αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα. Έχουμε συναντήσει πολλού stakeholders, πολλού εκπροσώπου από τον κλάδο αλλά και εκπροσώπου των κυβερνήσεων ε, και βρισκόμαστε σε επαφή και με όλου του σκιώδει εισηγητέ και τα διαφορετικά γραφεία των σκιώδων εισηγητών προκειμένου να φτάσουμε τελικά σε ένα συμβιβασμό στο πλαίσιο αυτού του αρκετά δύσκολου φακέλου. Και ταυτόχρονα ε, θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν θέλουμε να παρατήσουμε, ε, παρότι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε μια απάντηση σε αυτή την πρόταση τη Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σα παρουσιάσω ποιε είναι βασικέ αλλαγέ που προτείνουμε στο κείμενο τη Επιτροπή. Τι προτείνουμε δηλαδή από την πλευρά τη Επιτροπή μα. Καταρχήν, ε, τα όρια σε ό,τι αφορά ε, τις, ε, τις αποστάσεις προκειμένου να προστατευτούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Υπήρχε καταρχήν αυτό το όριο των 100 χιλιόμετρων από το οποίο και μετά, από την απόσταση δηλαδή αυτή και μετά, δεν μπορεί κανεί να παρεμποδίσει την είσοδο ενός μεταφορά σε άλλο κράτο μέλο. Εμεί εδώ έχουμε προτείνει κάποια ευαισθητότητα μέτρα, όπω για παράδειγμα στην τροπολογία 26. Δηλαδή, συμπληρωματικούς κανόνε που επιτρέπουν ακριβώ την παρεμπόδιση της εισόδου στην αγορά. Μία από αυτέ τι προποθέσει είναι ε, το αν, για παράδειγμα, υπονομεύει αυτό ο νέο παίκτη στην αγορά μια υφιστάμενη δημόσια υπηρεσία. Επίση, αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει με διαφανή τρόπο δυνατότητα επέκτασης αυτής, δηλαδή παρά παράταση τη υπηρεσία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχει νόημα ένα τέτοιο διαγωνισμό ε, σε σχέση με μια δημόσια ε, υπηρεσία που παρέχεται. Ε, μετά τίθεται και το ζήτημα των δρομολογίων που αποφέρουν κέρδη ή όχι, δηλαδή των κερδοφόρων. Οπότε ουσιαστικά εδώ θα πρέπει να υπάρχει λιγότερη επιβάλληση των φορολογούμενων και ε, περισσότερες διασυνοριακές ενισχύσεις όταν πράγματι υπάρχει κοινό όφελος διασυνοριακά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τα όρια. Από εκεί και μετά υπάρχει το ζήτημα της ε, ανάκληση αναστολή τη άδεια. Ε, προκειμένου να απευθυνθεί ε, η οποιαδήποτε καταστατήγηση αυτών των κανόνων σε ό,τι αφορά τι δημόσιε συμβάσει, ε, τα κράτη-μέλη με τη σύμφωνη γνώμη τη Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν ακόμα και να καλούν την άδεια σε ό,τι αφορά την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, εάν πράγματι το οικονομικό, η οικονομική ισορροπία σε ό,τι αφορά τι δημόσιε συμβάσει απειλείται. Και σε αυτή την περίπτωση δίνεται μια προθεσμία 6 μηνών στον ενδιαφερόμενο και αυτό το ζήτημα της οικονομικής ισορροπίας βέβαια συνδέεται ακόμα με κάποια ερωτηματικά, κάποιες εκκρεμότητες. Ε, γι' αυτό και αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί ότι δηλαδή κατά πόσο επαρκεί η χρήση ενός τέτοιου όρου απλώς και μόνο, δηλαδή του να λέμε ε, οικονομικό, οικονομική ισορροπία, οικονομικό ισοσύνη. Και μετά ε, επίσης αυτό που συμβαίνει είναι ότι τέτοιου είδους κανόνε ισχύουν σε διάφορου ε, τομεί. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τι δημόσιε επιχειρήσει κοινή ωφελία σε μία σειρά από, κράτα, από κράτη-μέλη. Ε, γιατί βέβαια ειδικότερα εδώ έχουμε να κάνουμε ε, με, με ρυθμιστικές αρχές ανεξάρτητες εδώ από την πλευρά των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για να προβαίνουν σε αυτή την χορήγηση όχι της άδειας τώρα. Μετά, περαιτέρω τροπολογίε έχουν να κάνουν ε, με τη δικαίωμα εξαίρεση ε, από το πεδίο εφαρμογή των αστικών περιοχών. Με άλλα λόγια, τι θέλουμε να πούμε. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά ε, την ειδική ρύθμιση σε ό,τι αφορά τις αστικές περιοχές. Γιατί η πρόταση εδώ στοχεύει στο να ανοίξει η αγορά σε υπεραστικό επίπεδο, αλλά όχι σε αστικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διατήρηση του συστήματο ε, στα κράτη-μέλη, χωρί να υπάρχουν ανησυχίε ω προ τι ε, αλλαγέ που θα μπορούσαν να προκύψουν σε αστικό επίπεδο. Επίση, κατά την συζήτηση που κάναμε με του ε, stakeholders, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε σε ό,τι αφορά τι καταχρήσει που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στην αγορά. Γι' αυτό στι τροπολογίε 3 και 28 ακριβώ προβλέπουμε κάποιε ρήτε για να αποφύγουμε την κατάχρηση τη αγορά. Προβλέπουμε δηλαδή ίσους ε, κανόνες ε, ε, του παιχνιδιού εντό εισαγωγικών που θα επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές της αγοράς σε ό,τι αφορά την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισέλθει για παράδειγμα κανείς στην αγορά με ζημία ε, ε, καταφέρνει να επιβληθεί στην αγορά ε, και μετά αυξάνει όσο θέλει τις τιμές. Θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε μια τέτοια κατάσταση και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση μέσω ακριβώς παροχής περισσότερων εξουσιών στις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να μην υπάρχει κατάχρηση αγοράς. Μετά, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους θεματικούς σταθμούς και το κατά πόσο θα αναφερόμαστε σε δημόσιου ή ιδιωτικούς, είπαμε τελικά ότι δεν θα γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα στου δημόσιου ιδιωτικού θεματικούς σταθμού, αλλά τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν κατά πόσο αυτοί οι τερματικοί σταθμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται μόνο από συγκεκριμένου μεταφορεί να είναι δυνατόν να περιορίζονται σε ό,τι αφορά τη χρήση του από όλου του μεταφορεί ή όχι. Ε, τώρα, ε, το ζήτημα της εγκατάστασης και η πρόταση που είχε γίνει από την Επιτροπή από την ένα ζήτημα δηλαδή είχε προταθεί από την Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο να εγγράφεται μια επιχείρηση η οποία αναλαμβάνει δραστηριότητα σε ένα άλλο κράτο μέλο. Ε, ωστόσο, τελικά αποφασίστηκε ότι εντό 6 μηνών θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι έχει πράγματι ο ε, συγκεκριμένο μεταφορέα εδρεωθεί σταθερά στον λόγο κράτο μέλο εντό 6 μηνών. Και από εκεί και μετά, δηλαδή μέσα σε αυτού του 6 πρώτου μήνε και μετά θα πρέπει να ε, εγγραφούν, να καταχωρηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά το καθεστώς που θα ισχύει, την, την ευελιξία δηλαδή που θα υπάρχει, προβλέπουμε να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη εκείνα που θέλουν να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ανοίγματο να το κάνουν. Ε, μετά, ε, Καταλήγοντα, αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα ακόμα αμφιλεγόμενο ζήτημα σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση. Ε, ε, και γνωρίζω πως υπάρχουν κάποιες φήμες ως προς τα προβλήματα ε, που θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτό το ζήτημα, αυτό ο φάκελος σε ό,τι αφορά το σύνολο του πρώτου πακέτου κινητικότητας, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει αυτό, γιατί ε, δεν ε, θα μπορούμε να εξηγήσουμε αν αποτύχουμε σε σχέση με αυτό στους πολίτες μας, στους ψηφοφόρους μας και ακόμα εδώ και στη Συμπρόεδρο το γιατί αποτύχαμε όταν αμοιβόμαστε τόσο άδρα να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζήλε για αυτή σας την εισήγηση εξήγηση πολύ σαφής και αρκετά διαφωτιστική για τις βασικές προκλήσεις του θέματος. Κύριε Ντεγκράντες Πασκουάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, Αντιπρόεδρε. Συμπρόεδρε της Επιτροπής Μεταφορών Καμίγη. Εντάξει το μικρόφωνο μου. Ε, να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας και εγώ αυτό που είπε ο συνάδελφος. Για την αναβολή τη όλη συζήτηση. Εάν πρέπει κάποιον να κατηγορήσουμε, δεν είμαστε εμεί. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθυστέρησε πάρα πολύ να υποβάλει τι σχετικέ προτάσει. Φέτο δεν έγινε τίποτα μέχρι τώρα. Εμένα δεν είναι ότι με πειράζει, αλλά τώρα μπορεί μόνο να αρχίσει να εργάζεται η Επιτροπή μα. Είναι δύσκολο λοιπόν να προλάβουμε να κάνουμε ό,τι και να χρειαστεί. Για τα θέματα των λεωφορείων και των πούλμαν. Ε, συνδέονται και με άλλα στοιχεία του πακέτου κινητικότητας. Οι σοσιαλιστές έχουν κάνει τις προτάσεις τους και γνωρίζω ότι θα μπορούσε η συζήτηση και λογικό θα ήταν να αναβληθεί. Καταλαβαίνω όμως και τον κύριο Ζήλε και όσα είπε στην παρέμβασή του. Έχουμε διαφορετικέ απόψει λοιπόν. Αυτό είναι σαφέ. Είναι περίπλοκο το θέμα και αυτό είναι σαφέ. Ο κύριο Ζήλε μα άκουσε στι συνεδρίε των ε, σχεδόν εισηγητών. Σημείωσε τι απόψει ε, των διάφορων συμμετεχόντων. Αλλά να είμαστε ειλικρινεί. Πολλέ από τι παρατηρήσει αυτέ απηχήθηκαν σε όσα μόλι μα είπε και στο κείμενό του και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλουμε να έχουμε μια έκθεση που να είναι σφαιρική, σφαιρικού περιεχομένου, να καλύπτει τις μέρημνες όλων. Να είναι καλό και για τα κρατημέλη, αλλά και για όσους θέλουν να διατηρήσουν τα κρατικά του συστήματα συγκοινωνιών. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να φροντίσουμε να ε, ικανοποιήσουμε και τις δύο πλευρές. Πάντως το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Είναι πολύ θετικό το κείμενο, πολύ ε, Για να μην επαναλάβουμε λοιπόν αυτό που μόλις είπε ο κύριος Ζήλια και που τα γνωρίζετε και πολύ καλά για το ισπανικό σύστημα, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Για τα χιλιόμετρα, η υποχρέωση της ε, δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό για μας ε, συμπίπτει με το ευρωπαϊκό καθήκον, ευρωπαϊκή υποχρέωση. Θα πρέπει εμείς συστηματικά να σεβόμαστε την ε, εξουσία που αναθέτουν τα κράτη-μέλη στους δημόσιους φορείς τους. Ο κύριος Ζήλε θέλει να προστατεύσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις κρατικές. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε τι προβλέπει και ο κανονισμός του 2007 που λέει ότι ε, τις αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά τις αναλαμβάνουν τα κρατημέλη. Με άλλα λόγια, πρέπει να κοιτάξουμε μήπως εδώ υπάρχει σύγκρουση με τις εθνικές αρμοδιότητες και το θέμα θα μπορούσε να έχει νομική, νομικές προεκτάσεις. Επίσης, θα θέλαμε να μην πάρει διαστάσεις δικαστικές το όλο θέμα, δηλαδή προσφυγέ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ούτω καθεξή. Το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή επιτρέπει ε, να καλλιεργούνται οι δημόσιες ε, μεταφορές που εργάζονται βάσει της αποκλειστικότητας. Δεν θέλουμε εδώ να δημιουργηθεί ένα νομικό μιλφέγι με διαφορετικές στρώσεις. θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ένα περιθώριο ελιγμού και να αποφασίζουν αν θέλουν να υπάρχει ανεξάρτητος ρυθμιστής ή όχι. Το καμποτάζ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δουν εάν ε, πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός ή όχι. Πρόεδρε, εδώ δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να αποφασίσουμε αν τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν τι αποφάσει μόνο του ή όχι. Και αν θα πετανεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο ή όχι. Και για το ισπανικό πρόβλημα, όπω ε, ονομάστηκε. Δεν είναι ισπανικό πρόβλημα. Είναι διαφορετικό το μοντέλο μας. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε την κερδοφορία τη χώρισης για να ε, χρηματοδοτήσουμε τι γραμμέ που δεν έχουν τέτοια κερδοφορία αλλά είναι κρατικέ ιδιοκτησία. Ιδάλω δεν θα μπορούσαμε να τι χρηματοδοτήσουμε, γι' αυτό έχουμε αυτό το σύστημα των εκχωρήσεων. Ε, δεν θα μπορούσαμε αλλιώ να χρηματοδοτήσουμε τι γραμμέ που δεν έχουν ιδιαίτερο κέρδο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η βιωσιμότητα ακριβώ και η διάρκεια ζωή του συστήματο ε, συγκοινωνιών μα. Τα πλεονεκτήματα του λεωφορείου και το πούλμαν είναι ότι επιτρέπουν την πρόσβαση που αλλιώ δεν θα συνδέονταν με άλλο μέσο. Δεν είναι λοιπόν ένα πρόβλημα αποκλειστικά ισπανικό. Ο κύριος Ζήλε ξέρει καλά ότι τα εθνικά κοινοβούλια της ε, Σλοβενία, τη Γερμανία, τη Γερμανίας, της ε, Αυστρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχίας έχουν αντιταχθεί στην πρόταση αυτή. Λέγοντα ότι προσβάλλεται η αρχή τη επικουρικότητα και τη ανάλογικότητα. Επίση, οι συνδικαλιστικέ οργανώσει των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών απέρριψαν την πρόταση. Γνωρίζεται λοιπόν τι συζητιέται στην Γερμανία, κυρίως για τους αστικούς και προαστιακούς, ε, τα αστικά και προαστιακά δίκτυα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις αντιρρήσεις και θα είμαι ειλικρινής και θετικός. Νομίζω ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα. Θα είναι δύσκολο να επιληφθεί και χρειαζόμαστε χρόνο κυρίως, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει άμεση σχέση με το πακέτο κινητικότητας και γνωρίζουμε ποιο ήταν, ποια ήταν ε, η τύχη του πακέτου αυτού και τι αντικσότητες πέρασε. Εγώ είμαι υπέρ της αναβολής όπως προτάθηκε από την ομάδα των σοσιαλιστών. Δεν είναι επί της ουσίας αντίρρηση. Ακόμη και αν υπάρχουν πολλά θέματα ουσία τα οποία έχουμε διαφορετικέ απόψει. Απλώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αναγκαίο να εμβαθύνουμε στο όλο θέμα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ο λόγο του κύριο Κουρούμπατσεφ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Αντέλη, νομίζω ότι θα ξεκινήσει 5.30 όπως είχε ανακοινωθεί η συζήτηση, γι' αυτό και έφτασα 5.30. Διαπίστωσα ότι είχε ξεκινήσει όμως ήδη ο εισηγητής, κατόπιν πήρε το λόγο η συνάδελφος Η πρόταση ουσιαστικά ξεκίνησε από την Επιτροπή. Ο κύριος Ζήλε, αξιοσέβαστος και έμπειρος συνάδελφος, προετοίμασε μια έκθεση. Αλλά όσον αφορά τη λογική της Επιτροπής, με το πακέτο 1 μας προτείνει περιορισμούς στο καμποτάζ. Από την άλλη, προτείνει για το εμπόριο αυτούς τους περιορισμούς και την ίδια ώρα για τους επιβάτες, για τη μεταφορά επιβατών, πλήρη απελευθέρωσε. Τελικά, με το καμποτάζ τι θα γίνει. Όπως είπα και σε μια πρώτη συζήτηση που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το καλό και το κακό καμποτάζ. Εγώ έχω μια εξήγηση. Όταν υπάρχει δεσπόδουσα θέση χώρας που ουσιαστικά βρίσκεται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, εκεί το καμποτάζ χαρακτηρίζεται κακό και θέλουμε να το περιορίσουμε. Όταν όμως δεσπόζουν δυτικής Ευρώπης επιχειρήσεις, ξαφνικά θέλουμε να συνεχιστεί η απελευθέρωση, γιατί είναι καλό το καμποτάζ. Η λογική μου είναι εντελώς διαφορετική όμως. Θεωρώ ότι στο εμπόριο μεταφορά φορτίων, εκεί βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει απελευθέρωση αντίθετα στις ε, μεταφορές επιβατών. Όταν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, έχουμε πάντα η δυνατότητα οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εγκατεστημένες ε, επιχειρήσεις να αντέξουν στην απελευθέρωση και να υπάρξει και μια μικρή προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κινδυνεύουν από πτώχευση και θα πρέπει να στηριχθούν είτε από τις κοινότητες, από τις περιφέρειες ή από τα κράτη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, επαναλαμβάνω τη λογική της Επιτροπής. Γιατί κάπου το καμποτάζ περιορίζεται και κάπου υπάρχει πλήρης απελευθέρωση. Επιπλέον, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποια εθνικά πρότυπα να εξάγονται αλλού. Αν είναι σωστό να εξάγουμε π.χ. το γερμανικό μοντέλο στην Ισπανία σε αυτή την περίπτωση το ισπανικό μοντέλο θα πρέπει επίσης να μπορεί να εξαχθεί στη Γερμανία. Και δεν είναι δουλειά ούτε της Επιτροπής, ούτε του Κοινοβουλίου να παίξει το ρόλο του εξαγωγέα ενός συστήματος από τη μία χώρα στην άλλη και στο τέλος να έχουμε το ίδιο πρότυπο και μοντέλο που να ισχύει παντού σε όλες τις χώρες. Γιατί αν μια μέρα επιβληθεί μία, αν θέλετε, και μοναδική λύση, θα δημιουργηθούν ενδεχομένως κοινωνικά προβλήματα παρόμοια σε όλες τις χώρες. Στη Γερμανία υπάρχει μονοπωλιακή κατάσταση και θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί αυτού του είδους το μονοπωλιακό μοντέλο είναι καλύτερο από το τοπικό. Ενδεχομένως με ένα τοπικό μοντέλο μεταφορών μπορεί κάποιος να έχει σαν συνομιλητή τον δήμαρχο ή τις ε, αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει συνομιλητής επιτόπου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει μία μοναδική απόφαση που να επιβληθεί και να εφαρμοστεί παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ικανοποιητικά σε μια χώρα, αλλού μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει, επαναλαμβάνω, ένα ενιαίο μοντέλο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές που οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι ουσιαστικά πρέπει να αποδείξουν στις ρυθμιστικές αρχές την οικονομική τους βιωσιμότητα και ισορροπία. Προς το παρόν, δεν υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις ε, όταν ας πούμε οι δημόσιες μεταφορές ε, γίνονται δωρεάν καμία οικονομική βιωσιμότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε πολλές αστικές μεταφορές, συγκοινωνίες, δεν μπορεί να επιβιώσουν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις, τα δημόσια μέσα μεταφορών όταν θα πρέπει να εξεταστούν, η βιωσιμότητά τους να εξεταστεί από έναν ε, ρυθμιστικό φορέα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί με αυτόν τον τρόπο θα επιβάλλουμε, όπως κάναμε και με τους οδηγούς φορτηγών, τις ίδιες επιβαρύνσεις και για τους οδηγούς των λεωφορείων και των πούλμαν. Πραγματικά αναρωτιέμαι όταν μιλάμε για καμποτάζ, όταν μιλάμε για αποσπασμένους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι κανόνες, ίδιοι κανόνες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες σε αυτού του είδους τις μεταφορές, να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε σε όλες τις μεταφορές τους ίδιους κανόνες. Θα υπάρξουν λοιπόν πάρα πολλές τροπολογίες και σε γενικές γραμμές δεν νομίζω ότι θα στηρίξουμε τον εισηγητή, ο οποίος ουσιαστικά σε γενικές γραμμές στηρίζει την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε λίγο να συντομεύουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Ρικέ, έχετε το λόγο. Πώς να είμαι σύντομος, είναι περίπλοκο το θέμα. Η επικουρικότητα εδώ είναι μέσα ε, μπροστά μας ακριβώς γιατί είναι η εθνική πραγματικότητα το σημαντικότερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, συγχαίρω τον Ρόμπερτ γιατί έκανε κάτι που δεν είναι εύκολο προσπαθώντα να καταλήξει σε μια έκθεση με τι εργασίε όλων των σχεδόν εισηγητών. Όμω, νομίζω ότι κατάλαβε ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Υπάρχουν ε, παγίδε Γι' αυτό το επεξεργαστήκαμε τόσο προσεκτικά πριν φτάσουμε ως εδώ. Αυτό που άκουσα από τους προηγούμενους και οδησυγητές είναι ότι τα μοντέλα είναι εξαιρετικά διαφορετικά. Για λόγους, ιστορίες και γεωγραφίες απλούστατα. Στις μικρές χώρες. Γεωγραφικά μιλάω για τις διαστάσεις. Ε, τις επιφάνειες. Ε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά από τι χώρε με μεγαλύτερη επιφάνεια. Κάποιε ε, χώρε έχουν σιδηροδρομικό δίκτυο, οπότε δεν έχουν την ίδια ιστορία και ίδια ανάγκη μεταφορά επιβατών οδικό. Εάν δούμε χώρε με υποδομέ σιδηροδρομικέ που δεν είναι πολύ πυκνό το δίκτυό του, εκεί είναι πολύ πιο σημαντικέ ε, οι οδικέ μεταφορέ για τη μεταφορά των επιβατών. Ενώ το αντίστροφο επίση ισχύει. Δεν είναι τα ίδια τα προβλήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει λοιπόν ε, σαφής ε, σχέση με την επικουρικότητα. Μετά το θέμα είναι και τα όρια εδώ, τα τα όρια. Το όριο των 100 χιλιόμετρων που αναφέρεται ας πούμε. 100 χιλιόμετρα στο Βέλγιο είναι φοβερό και στην Ισπανία είναι πολύ λιγότερο. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα όριο που θα εφαρμόζεται ομοιομόρφως σε όλη την Ευρώπη. Ένα δεύτερο σημείο για τα όρια, που μου φαίνεται πολύ περίπλοκο, είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να ακουμπήσουμε τους αστικού, τις αστικές ε, μεταφορές, αλλά μεταξύ των αστικών, των προαστιακών, τα περιφερειακά και ε, όλων των υπόλοιπων υπάρχουν ε, και οι περιφερειακοί, που αρχίζουν και που τελειώνουν τα όρια αυτά, γιατί όλα εξαρτώνται από το κάθε αστικό κέντρο. Ε, διότι κάθε φορά ο περιφερειακός ξεπερνάει λίγο τα όρια του αστικού κέντρου χωρίς να πηγαίνει πολύ μακριά. Άρα υπάρχει πρόβλημα του πώς ορίζει ο καθένας το περιφερειακό. Κάποιοι είναι ιδιοκτήτε, κάποιοι όχι και τελικά επιβαρύνεται ιδιοκτήτε για τι δραστηριότητε άλλων που απλώ έχουν πάρει την έγκριση. Για το καμποτάζ. Άκουσα τι παρατηρήσει του προηγούμενου συναδέλφου, μίλησε για το καμποτάζ και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα του πω κάτι το απλό. Δεν υπάρχει καμποτάζ για τα εμπορεύματα και καμποτάζ για του επιβάτε. Υπάρχει καλό και κακό καμποτάζ. Ε, το καμποτάζ για τα εμπορεύματα και του επιβάτε, το μόνο που επιδιώκει είναι η βελτιστοποίηση ας πούμε των διεθνών μεταφορών. Το κακό καμποτάζ είναι το καμποτάζ που γίνεται δραστηριότητα που ε, είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Αυτό βλέπουμε στα εμπορεύματα, αλλά συνήθω δεν συμβαίνει στι ε, μεταφορέ των επιβατών. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, υπάρχει το καλό και το κακό καμποτάζ. Υπάρχει το καμποτάζ που σκοπό έχει να αποφύγει να γυρίσει κάποιο άδειο. Υπάρχει το καμποτάζ που σκοπό έχει κάτι άλλο. Πάντω, σαφώ, αν γίνει μία δραστηριότητα που είναι αυτό σκοπό, είναι κακό καμποτάζ. Για τι υπηρεσίε του επιβάτε, το ίδιο δεν είναι το ίδιο να μεταφέρει κανεί κυβότια ή να μεταφέρει επιβάτε βεβαίω. Προφανώ υπάρχουν άλλοι κανόνε που να ισχύουν ανάλογα με τι υπηρεσίε που θα πρέπει να προσφέρουν. Δεν θα μακρηγορήσω. Είπατε, Πρόεδρε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αυτό που βλέπω είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει πειρασμός, δεν λέω απόπειρα, πειρασμός να το υπονομεύσουμε το θέμα αυτό και λόγω του, της ουσίας του περιεχομένου. Και για καλούς και για κακούς λόγους. Οι καλοί λόγοι είναι ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τις εθνικές αρμοδιότητες, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα το αποδείξει ως και η περαιτέρω συζήτηση. Ο, οι κακοί λόγοι είναι να αποφύγουμε το να συζητηθεί το θέμα και κατά συνέπεια να γίνει η ε, με διαφορετικούς υπόγειους τρόπους η καταβήθηση του όλου θέματος. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Κύριε Κράμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ συχνά τον, ε, θερμά τον Ρόμπερτ για, την, για αυτό το πρώτο σχέδιο και φυσικά πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα. Η Επιτροπή έχοντας κάνει την πρότασή της είτε την έκανε καθυστερημένα ή δεν έχει λάβει υπόψη της ε, τις ε, νέες εξελίξεις. Είναι σαν να παίρνει ως πρότυπο το γερμανικό μοντέλο. Και θα μπορούσε κανείς ε, να το πει αυτό πριν από τέσσερα χρόνια, ότι δηλαδή άνοιξε αγορά, υπήρξε πολλή ανταγωνισμό, πολλοί ανταγωνιστές και όλα αυτά ήταν ελκυστικά. Αλλά ήδη από τότε δεν θεωρούσα ότι έγινε κάτι εναντίον του αθέμητου ανταγωνισμού. Γιατί, για παράδειγμα, τα επεραστικά ε, δεν χρειάζονται να πληρώνονται διόδια, αλλά άλλε μεταφορέ δεν χρειάζεται να πληρώνουν διόδια. Και το ότι δεν θίγεται καν αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Γιατί δεν μπορεί να θεωρείται αυτό θεμητό ανταγωνισμό. Και ένα δεύτερο ζήτημα, όταν τελικά υπέβαλε την πρόταση τη Επιτροπή, η κατάσταση στη Γερμανία έχει αλλάξει τόσο πολύ έτσι ώστε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για μονοπόλιο στη Γερμανία. Και δεν γνωρίζω, δεν, δεν ήξερα ότι η Επιτροπή τάσεται υπέρ του μονοπωλίου. Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή είναι υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάσταση στη Γερμανία ως κατάσταση ελεύθερου ανταγωνισμού. Ουσιαστικά δηλαδή όσοι έχουν παραμείνει έχουν εξαγοράσει όσους ανταγωνιστές είχαν ε, μείνει στην αγορά με αποτέλεσμα να έχει μείνει ένας, να έχει μείνει ένα μονοπόλιο και δεν μπορεί αυτό να αποτελεί το υπόδειγμα για το υπόλοιπο της Ευρώπης από την άλλη πλευρά τώρα ε, κάναμε διάφορες συνομιλίες, για παράδειγμα και ειδικότερα με την Ισπανία, όπου η Ισπανική αγορά λειτουργεί πραγματικά εύρημα χωρίς να υπάρχουν, υπάρχει μονοπόλιο και όπου υπάρχουν ε, διάφοροι ανταγωνιστέ. Μου είπαν, για παράδειγμα, ότι 230 επιχειρήσει ε, δραστηριοποιούνται εκεί. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιηθεί το ισπανικό μοντέλο για τα υπεραστικά ε, λεωφορεία, για τα και γιατί δεν προσπαθεί να κάνει μια διόρθωση σε ό,τι αφορά αυτή την προσέγγιση. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι αυτές οι μεταφορές ε, ε, κοντινών αποστάσεων δεν θα πρέπει να ε, υπονομευτούν. Αλλά σας λέω, αυτές οι επιχειρήσεις καταβάλουν διόδια, αλλά όταν έρχομαι σε επαφή με τους ε, ε, διαχειριστέ των υπεραστικών ε, μα λένε ότι αφού δεν πληρώνουν διόδια οι PSO δεν θα πρέπει να πληρώνουμε κι εμεί. Μα αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ε, εντάξει, σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε τις μεταφορέ <clears throat> μεταφορές κοντινών αποστάσεων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ελεύθερο ανταγωνισμό. Και σα λέω από δική μου εμπειρία στη Γερμανία δεν λειτουργούν καλά τα, ε, τα πράγματα, δηλαδή δεν θέλουμε μονοπόλιο όπως αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει στη Γερμανία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τέρμινα στου θερματικού σταθμούς, τα πράγματα είναι περίπλοκα. Εάν κατασκευάσουμε ένα τερματικό σταθμό με δημόσια χρήματα, με δημόσιο χρήμα, δεν μπορούμε να το διαθέσουμε σε έναν και μόνο μεταφορέα αλλά όταν έχουμε να κάνουμε ε, με ιδιωτικό μεταφορείο ο οποίο έχει κατασκευάσει ένα δικό του τερματικό σταθμό, τι θα κάνουμε, θα τον υποχρεώσουμε να καταστήσει διαθέσιμο αυτόν τον τερματικό σταθμό σε άλλους ε, μεταφορεί. δεν έχει αυτό νόημα. Οπότε δεν νομίζω πω το έχει σκεφτεί καλά αυτό το σύστημα η Επιτροπή που θέλει να δημιουργήσει. Και από εκεί και μετά βέβαια χρειαζόμαστε και ασφάλεια δικαίου. Υπάρχουν λοιπόν παραδείγματα τα οποία μπορούν να μα βοηθήσουν στους σιδηροδρόμους όπου αποφύγαμε το cherry picking, δηλαδή να ε, επιλέγει κανείς μόνο τις ε, δίδαξη που επιθυμεί για παράδειγμα. Έγινε ένα ε, διαγωνισμό σε συγκεκριμένη πόλη της Γερμανίας, τέσσερις είχαν ενδιαφερόμενοι και επιλέχθηκαν δύο. Και είπαμε, σε ό,τι αφορά τι προσφορές που είχαν υποβληθεί, η κινητικότητα θα πρέπει να είναι η βασική μα αρχή. Και κατά συνέπεια, ε, για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές ε, εγώ ε, μπορώ να βγάλω πολλά, ταυτόχρονα θα πρέπει να εξυπηρετήσω και τις λιγότερο, τις πιο αραιοκατοικημένες περιοχές. Πρόεδρε, μου λέτε να μιλήσω πιο, να, να, να συντομεύσω, αλλά οι προηγούμενοι δύο μιλητέ μακρηγόρησαν πάρα πολύ, οπότε θα ήθελα και εγώ να μιλήσω. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι σε αυτόν τον τομέα χρειαζόμαστε θεμετό ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. La Ευχαριστούμε, κυρία Βιού. Ναι, ο συνάδελφός μου Ζωάο Πιμέντα Λόπε, έχει μείνει στην Πορτογαλία και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ. Ευχαριστεί τον ε, εισηγητή και θα ήθελε να διαβάσω τι παρατηρήσει του για την έκθεση αυτή ως σκόπος εισηγητή για την ΚΟΕ. Η πρόταση αυτή ε, ανήκει σε μια προσπάθεια απελευθέρωση του τομέα των συγκοινωνιών για να διευκολυνθεί η είσοδο των πολυεθνικών εταιριών στον χώρο τη αγορά της εθνικής και να δημιουργηθούν να αποδομηθούν τα εργαλεία που μέχρι τώρα επέτρεπαν στα κράτη-μέλη να ρυθμίζουν τον όλο κλάδο στη δική του επικράτεια και να αποφασίζουν πώ θα γίνεται η εμπορία στη δική του αγορά και μεταφορά των δικών του επιβατών. Μα λένε ότι είναι για να αποφύγουμε το υπερβολικό διοικητικό άχθο για την ε, ε, έλευση στην αγορά. Στην πραγματικότητα όμω αυξάνεται το κόστο για τι αστικέ και προαστιακές κοινωνίε. Διευκολύνεται η καμποτάζ, η χρήση λεωφορείων και πούλμαν άλλων κρατών μελών στα εθνικά δίκτυα μια χώρας και ε, τίθενται εν κινδύνο τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, πλήττεται επίσης το εργατικό δίκαιο εκεί όπου οι ε, κανόνες και οι μισθοί είναι πιο υψηλοί. Για τα τερματικά και τους σταθμούς, με την ίδια κριτική πρόσβαση στα τερματικά. Ουσιαστικά δίνεται προτεραιότητα σε μια ιδιαίτερη μορφή υποδομών για να ευνοηθούν όχι οι εθνικές εταιρείε, αλλά οι ε, επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να πάρουν μια παραχώρηση για την λειτουργία αυτού του τερματικού. Αυτές όμως οι εγκαταστάσεις συνήθως κατασκευάζονται με δημόσιο χρήμα, με δημόσιε επενδύσει. Πρόκειται για επεξαίρεση στην πραγματικότητα των δημοσίων, δημοσίων κονδυλίων προ όφελο των ιδιωτών, ιδίω των μεγάλων ομίλων, χωρί να έχει δυνατότητα ο δημόσιο τομέα να πάρει το κέρδο αυτών των επενδύσεων. Ω προ τι διαδικασίε των διαβουλεύσεων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όσων αγωνίζονται για να προασπιστούν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Γι' αυτό θα υποβληθούν τροπολογίες από το Ζωάο Πιμέντα, που είναι ο σκιώδης συζητητής, για να προασπιστεί τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις δημόσιες επενδύσεις προς όφελος των πολιτών και του λαού, και για να έρθει αντιμέτωπος με την απόλυτη απορρίθμιση προστατεύοντα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ευχαριστούμε κυρία Βιού. Κυρία Άντερσον, εσείς τώρα. Και μετά θα ολοκληρώσουμε την κυρία Ντεμόντε. Α, και η κυρία Γιάλα Ζέντερ. Θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί πολλά από αυτά που ήθελα να πω ακούστηκαν ήδη. Συμφωνώ με τον κύριο Τικλάντες και τον κύριο Κρόμπαχερ. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό πίσω από αυτή την πρόταση και πιστεύω ότι θα στοχεύσουμε πολύ περισσότερο το Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο μήνα, στο δείπνο που είχαμε με τους συνδικαλιστές, της Δημοσίας αρχές, τους εμπλεκόμενους φορείς, εκπροσώπους του Συμβουλίου και πάρα πολύ λίγοι είχαν να πούν κάτι καλό για αυτή την πρόταση. Ακούσαμε τον επικεφαλής της DigiMove που μα την παρουσίασε την πρόταση και ακούσαμε πολύ προσεκτικά αυτά που ήθελε να μα παρουσιάσει. Κάναμε συγκεκριμένε παρατηρήσει. Υπάρχουν προβλήματα και όσον αφορά τη μέθοδο και βλέπουμε πίσω από αυτή την πρόταση την ενίσχυση των διεθνών ουσιαστικά επιχειρήσεων και ομίλων και φορέων. Αυτού στηρίζει η πρόταση αυτή και όχι τους ε, φορείς εντός της Ευρώπης, ούτε τους εθνικούς και τοπικούς. Βλέπουμε ότι μόνο κάποιοι από τους φορείς έχουν εισακουστεί δεν υπάρχει απολύτως ε, κανένα στοιχείο που να έχει συγκριθεί. Είναι ουσιαστικά σαν να αλλάζουμε πρότυπο ξαφνικά. Γιατί είναι καλύτερα τα λεωφορεία σε σχέση με τα γιοταχή. Πλήττουν λιγότερο το περιβάλλον, όπως είπε ο κύριος Κράμπερ, είναι σωστό σε σχέση με το κατακεφαλήν, αν θέλετε, τε, ε, κόστος, αλλά και το κατά πόσο πλήττεται το περιβάλλον, το τοπίο. Ο κύριος Ζήλε προσπάθησε με τις τροπολογίες να λάβει υπόψη τους αυτή την πτυχή. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ε, ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες ε, αρχές στα κράτη-μέλη μας σε σχέση με την πυκνότητα κατήχησης κάποιων περιοχών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Ντεμόντα, ευχαριστώ πρόεδρε. Χαιρετίζω και την αντιπρόεδρό μας. Ε, καλή τύχη στις εργασίες σας. Μια πολύ σύντομη παρέμβαση για να αναφέρω και εγώ τις δικές μου παρατηρήσεις, ευχαριστώντας τον γιατί και τους κοιόδης για τις παρεμβάσεις τους. Αποσαφενίστηκαν κάποια πράγματα. Όμως, να πω ότι απελευθερώνοντας την αγορά, δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει σίγουρα ο κλάδο των μεταφορών στην Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστικό ε, και πιο αποτελεσματικό, αλλά να δούμε και τι εναλλακτικέ έχουμε στι μεταφορέ. Διότι ω προ τα καθαρά ενεργειακώ οχήματα, θα πρέπει ίσω να παροτρύνουμε στη χρήση των σιδηροδρόμων ή να υπάρχει ε, κοινή χρήση των διτρόχων ε, ή των ιδιωτικών οχημάτων. Ε, είναι ένας τρόπος λοιπόν και το τα λεωφορεία για τα πούλμαν. Ε, τώρα για το καμποτάζ θα πρέπει να δούμε πώς θα διευθετηθούν αυτά και να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες και για τα εμπορεύματα και για τα λεωφορεία, δηλαδή τη μεταφορά επιβατών. Θα πρέπει σίγουρα να είναι ομοιόμορφη η αντιμετώπιση και από το καμποτάζ ε, να κοιτάζουμε, να, να πατάσουμε το ανεξέλεγκτο καμποτάζ. Υπάρχει και μια μορφή υγιής και υπάρχει και το θέμα του ανοίγματο της αγοράς. Νομίζω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις συμβάσεις κοινή ωφελία, τι δημόσιε συμβάσει και μια τελευταία κουβέντα για την ασφάλεια. Βεβαίω είναι διαφορετικά πράγματα η μεταφορά ανθρώπων και πολιτών και η μεταφορά εμπορευμάτων. στη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν κάποιο μεταφέρει 30 τόνου, αυτό από μόνο του αποτελεί κίνδυνο. Ε, δεν είναι το τι εμπόρευμα είναι. Είναι ότι 30 τόνοι στους δρόμους είναι ένας κίνδυνος. Θα πρέπει λοιπόν πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ε, αυτούς τους κινδύνους και να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί με τέτοια φορτία που μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Θα είναι ένας σοβαρός κίνδυνος και θέλουμε στους δρόμους να υπάρχει ασφάλεια. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε, κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Δεγκράντες και με τον συνάδελφο Κορόμ Μπάτσεφ. Πράγματι, νομίζω ότι το ισπανικό μοντέλο δεν είναι καλύτερο ούτε χειρότερο από άλλα. Απλώς κατανοώ γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιζητά τρόπους προστασίας. Ξέρετε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε. Ε, και ξέρουμε τι συμβαίνει όταν δεν προβλέπεται προστασία, όταν υπάρχουν διαγωνισμοί που είναι τελείως ανοιχτοί. Λέτε ότι στην Ισπανία δεν έχουμε προβλήματα, όμως με περίπλοκη γεωμορφολογία, ε, με χωριά που είναι τελείως απομονωμένα, παρόλα αυτά το σύστημα λειτουργεί. Πολλές φορές χρειάζεται να τετραγωνίσουμε τον κύκλο για να βρούμε τρόπους να παρέχονται υπηρεσίες μεταφορές στο σύνολο της επικράτειας, στο σύνολο της επιφάνειας και σε όλη τη γραμμή. Όχι μόνο για κάποιο μέρος κάποιας γραμμής, για το σύνολο του δικτύου. Ε, ε, Βεβαίω λειτουργεί καλά το δίκτυό μα, αλλά θέλουμε και ένα νέο του στόλου, ε, θέλουμε καλύτερα οχήματα, θέλουμε περισσότερη ασφάλεια για του επιβάτε. Και αυτή τη στιγμή περνάμε μια κρίση τρομερή. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε και το σωστό σημείο ισορροπία. Από την άποψη των ε, επενδύσεων, την άποψη τη χρηματοδότηση. Προκειμένου οι κρατικέ αρχέ που ε, τις ελέγχουν οι ευρωπαϊκές με τη σειρά τους για τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να καταφέρουν να παρουσιάσουν κάποια κερδοφορία. Νομίζω ότι απλώς το γεγονός ότι πληρώνονται ε, ε, στις εταιρείες κάποιες κρατικές βοήθειες είναι ένας καλός τρόπος. θα έρθουν εκλογέ. Μην κοιτάξουμε να αποσαρθρώσουμε ή να καταστρέψουμε συστήματα που λειτουργούν καλά. Νομίζω ότι ακόμη και στους διαγωνισμούς υπάρχουν ξένες εταιρείε, ε, παίρνουν μέρος ξένες εταιρείε. Και παρέχουν ε, υπηρεσίε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά διακριτική μεταχείριση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το κοινοβούλιο μα να κάνει ό,τι μπορεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην επιδεινωθεί η κατάσταση σε ένα σύστημα που είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και σε κάποιε χώρε λειτουργεί καλά. Γεωγραφικώ δεν είναι απλό να παρέχουμε υπηρεσίε μεταφορών σε όλη την Ισπανία. Ε, νομίζω ότι το σύστημα επεβίωσε τι κρίση. οι χρήστε είναι ικανοποιημένοι και καλό θα ήταν να δούμε ε, τι θέλουμε για το μέλλον. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ, να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ράσμουσεν. Θα σας παρακαλέσω να είστε συνοπτικότατος. Ευχαριστώ Πρόεδρε για όλα τα σχόλια και ειδικότερα του κύριου Ζήτη για αυτήν την ε, έκθεση που θεωρούμε πως οι γενικές γραμμές υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής. Επιτρέψτε μου να σας επενθυμίσω πολύ ε, σύντομα τον στόχο της πρότασης της Επιτροπής. Είναι ε, να δούμε το το νέο μοντέλο το οποίο επιβάλλεται ε, σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο των ε, λεωφορείων και πούλμαν και ε, θεωρούμε πως οι βελτιωμένες υπηρεσίες λοιπόν σε αυτό το τομέα θα αποτελέσουν μια βελτίωση και της ανταγωνιστικότητας σε αυτό το τομέα και θα ενισχύσουν την κινητικότητα των πολιτών, ειδικότερα πολιτών οι οποίοι δεν έχουν άλλη δυνατότητα να μετακινηθούν όπως έχει καταδείξει και μια πρόσφατη γαλλική μελέτη. Αυτοί λοιπόν είναι οι επιβάτες τους οποίους ε, εστιάζουμε ιδιαίτερα. Ε, οι περισσότερες από ε, του κυρίου Ζήλε από τη δική μας πλευρά θεωρούνται πολύ θετικές και σε ό,τι αφορά την προστασία των δημοσίων συμβάσεων εδώ πράγματι είναι πολύ σημαντική και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αρνούνται τέτοιου είδου ε, παροχή υπηρεσιών ανάλογα ε, με το ε, τι νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Και επίση ο εισηγητή προτείνει μια τροπολογία η οποία θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να, να λάβουν συμπληρωματικά μέτρα εάν η παροχή ακριβώς εκτέλεση μιας δημόσιας υπηρεσίας θα είχε, θα επιδεινωνόταν από την ε, είσοδο στην αγορά ενός τέτοιου νέου μεταφορέα. Και επίσης ε, ε, ε αναφέρεται σε αυτή την τροπολογία ότι θα μπορεί να γίνεται μια άρνηση σε ό,τι αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα. Πράγματι αυτά τα θεωρούμε σε θετικές τροπολογίες για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης ο εισηγητή ε, προτείνει ένα μέτρο το οποίο θα επιβάλλει στου μεταφορείς να συμμορφώνονται με, τις, ε, με τους κανόνες της εγκατάστασης που ισχύουν στο κάθε κράτο μέλο. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η προϋπόθεση ε, θα πρέπει να πληρεί ορισμένε προποθέσει έτσι ώστε να μην οδηγήσει ουσιαστικά στην, στην δυσκολία εισόδου μέσα σε μια εθνική αγορά. Σε ό,τι αφορά του τομεί στους οποίου θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά είναι ο ορισμό των τερματικών σταθμών, των Τερμινάλ, για το γεγονό ότι θα πρέπει να εγκρίνονται προτούν χαρακτηριστούν ως τερματική ε, σταθμή αυτά τα terminals, ίσως να οδηγήσει στο πρόβλημα στο να, στο να μην περιληφθούν πλέον στο πεδίο εφαρμογή μια σειρά από τερματική σταθμή. Σας ευχαριστώ πολύ και να κάνω και ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την επιβολή των τελών. Ε, θα θυμόσαστε πω την ε, πρόταση τη Επιτροπή που είχαμε κάνει σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σήμα Τέλου Κυκλοφορία, τη Βινιέτα, είχαμε συμπεριλάβει και τα λεωφορεία και τα πούλμαν ή τα υπεραστικά λεωφορεία. Και ε, πράγματι προτείνουμε λοιπόν να περιληφθούν εδώ στην, ε, στο πεδίο εφαρμογή του, ώστε να έχουμε ναι, θεμητό ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Θες να τα πεις στη μαμά σου, ε. ε ο κύριος Ζήλε, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι για αυτή την τόσο ειλικρινή και έντιμη ανταλλαγή απόψεων. Δύο παρατηρήσεις για να ξεκαθαρίσω. Δεν προτείνουμε μόνο την απόσταση και τα 100 χιλιόμετρα, αλλά τέσσερα ακόμη κριτήρια τα οποία θα συμπεριληφθούν σε τροπολογίες, τα οποία θα επιτρέπουν σε, μια, ε, ε, σε ένα κατοσμέλος να μην ανοίξει την αγορά για το πάνω από τα 100 χιλιόμετρα, για τους φραγμούς, και τις μοιαστικές συγκοινωνίες το Τάλιν μπορεί να το κάνει όπω θέλει. Ο δήμαρχό του μπορεί να κάνει αυτό που έκανα και εγώ αν είναι τόσο έξυπνο. Για του σιδηροδρόμου. πολλά μέρη που κατοικούνται αεροκατοικημένα δεν συνδέονται με σιδηροδρόμου. Κάποιε φορέ ε, θα πρέπει κανεί να διανύσει 100 χιλιόμετρα με ποδήλατο. Δεν γίνεται. Ποιο μπορεί να κάνει 100 χιλιόμετρα με ποδήλατο. Εγώ μπορώ. Θα τα κατάφερνα, αλλά πολλοί άλλοι όχι. Συνάδελφοι, στην επιχειρηματολογία μας παρακαλώ να είμαστε σοβαροί και σε γενικές γραμμές για την ενιαία, για την ενιαία αγορά πιστεύω στο μέλλον θα πρέπει να ξερούμε το καμποτάζ. Δεν μπορεί να έχουμε ενιαία αγορά και να υπάρχει καμποτάζ. Οικονομικός μιλώντας. Πάντως αυτό είναι το πολύ μακρινό μέλλον. Ε, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι με πολύ μικρά βήματα σιγά σιγά μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία ανταγωνισμού. Εγώ πιστεύω στον ανταγωνισμό και λέμε διαρκώ θέλουμε στενότερη ένωση, περισσότερη Ευρώπη, τόσο το καλύτερο. Ε, η Ευρώπη είναι μια νέα αγορά με ελεύθερε υπηρεσίε. Αλλιώ πώ είναι στενότερη και περισσότερη Ευρώπη. Και από πολιτική απόψη να είμαστε λίγο συνεπεί με την ορολογία μας και με τις απόψεις μας. Ε, ευχαριστώ πολύ και στο μέλλον σκοπεύω να συνεργαστώ ε, επικοδομητικά με όλους τους συναδέλφους. Παρακαλώ υποβάλλετε τις τροπολογίες σας για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστούμε κύριε Ζήλε. Η υποβολή τροπολογιών και η προθεσμία τους λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Και πριν φύγετε η συμπρόεδρός μου έχει δύο κουβέντες να σας πει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βοηθεί γραμματεία και διερμηνείς. Θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους. Καλές διακοπές. Ζήτω η Γαλλία, ζήτω η ομάδα του Βαλγίου. Πρόεδρος, όλοι θα κερδίσουμε σήμερα το βράδυ. Σας καλώ όλους στον τρίτο όροφο. Σας εύχομαι καλές διακοπές ξεκούραστες. Κύριε Πασκουάλ, έχετε το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την μικρή μας αντιπρόεδρο, η οποία μιλάει πάρα πολύ ωραία. Κάναμε μία πρόταση, ανεπίσημα εγώ, αλλά και επίσημα κάποια άλλη. Η πολύ αυτή της έκθεσης και η αλλαγή όσον αφορά την ημερομηνία. Ναι, διαφωνεί, φαντάζομαι, ο εισηγητή. Μήπω όμως πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Είναι ναι. στην ημερήσια διάταξη, θα το σκεφτείτε. Κύριε Ντεγκράντες. δεν σκέφτομαι από εδώ και πέρα, γιατί ξεκινάνε οι διακοπές μου και θεωρώ ότι το σημείο αυτό θα μπει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης των εισηγητών, καθότι οι εισηγητές θα πάρουν την απόφαση αυτή. Φυσικά και δεν σταματάω να σκέφτομαι. Εγώ θα συνεχίσω και την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πακέτο για την κινητικότητα. Καλούμε και τους διερμηνείς στο τρίτο όροφο. Ελάτε να πάρετε ένα φωτό μαζί μας. Καλές διακουπές σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκουραστείτε στον ήλιο, στη θάλασσα, στην εξοχή.